ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και λαμβάνω υπόψη και την ψήφο του κυρίου Σιλβέστρης. Εγκρίνεται. Άλλωστε τώρα έχει διορθωθεί και η συσκευή του. Τροπολογία 84, ο Λενίτσακ. Ποιος είναι υπέρ, διανατάσσου της χειρός παρακαλώ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 83, Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 83 του κυρίου Γιάρ άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας ισοπαλία απορρίπτεται 85 Έλγορτ σηκώστε τα χέρια παρακαλώ 85 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 σε και ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 Φερέιρα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 89. Νικουλέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την τροπολογία 89. Νικουλέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90 τώρα. Σηκώστε τα χέρια, Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99, Γκάμπριελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 92, Φερέιρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 93, Γκάμπριελ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 Άιλουρτ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 Σιλβέστρης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99. δαντσίλα, Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 το κυρίου Σεκέρς και του εισηγητού ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 Σιλβέστρης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 Λιούπτσεβα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 103 Φερέιρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 Ντόρφμαν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 Νικουλέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 Νικουλέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 Σάρμπου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 Φερέιρα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 Γέαρ υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 112 του κ. Πέτερ Γιάρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 113. Ψηλά τα χέρια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 114 άλβες υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 114 του κ. Άλβες άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 114 του κ. Άλβες με μεγάλη διαφορά Διανατάσσεως της χειρός. 115. Φερέιρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Ντάντσιλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται. 118. Του κυρίου Γιάρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μάλλον. 117. Ντόρφμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 λέει ο πρόεδρος. συγγνώμη, οι τροπολογίες 119 και 120 έχουν αποσυρθεί. Περνάμε στην 121 λέει Αρίκ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5. Γκαρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 Λιαρίκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 Φερέιρα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, Λιούπτσεβα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, Μπαράτσου, υπέρ, διανατάσεις της χειρός, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται, τι λέτε. Ζωζέσικ, κάνε τον έλεγχο. Τροπολογία 12, Βοητσεχόφσκι, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Γέγκλε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 14. Μπαράτσου. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 15. Λεϊαρίκ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Βοητσεχόφσκι. Υπέρ. Κατά Αποχέ, Μάλλον εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Aylward. Α, όχι, έχει διαγραφεί. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε παρόλα αυτά. 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Ντόρφμαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18 του κυρίου Ντόρφμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione ηλεκτρονικά κιούσα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 18 του κυρίου Ντόρφμαν. Προχωράμε στην 20. Λεϊαρίκ. Διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Σάρμπου υπέρ. Κατά δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 21, Λιαρίκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α, όχι, λάθος, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Φερέιρα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, Aylward, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26, Γιάρ. ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27, ε, ή μάλλον όχι, 29, 27 καταπίπτει. 29, Φερέιρα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 του κυρίου Σεκέσκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 άλβες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 Ντόρφμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Σάρμπου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Ρόντουστ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 36 της κυρίας Ρόντουστ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 35 Aylward. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 Μπαράτσου. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές μάλλον εγκρίνεται. περίεργο. Γιατί πρόκειται για ε, τροπολογία της συναδέλφου από σοσιαλιστές και δημοκράτες και βλέπω ότι το, η ομάδα της καταψηφίζει. Ας το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 38 Μπαράτσου. Αυτές είναι οι αλχημίες της πολιτικής. Τροπολογία 39 Σάρμπου, διανατάσεις χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, Φεραίρα και πάλι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συνεχίζουμε 46 ντάντσιλα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 ντάντσιλα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 γιάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 Βοητσεχόφσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 Σάρμπου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 Λιαρίκ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 55 Γκάμπριελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το ούτω τροποποιηθέν ψήφισμα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Συγχαρητήρια στον κύριο Σεκέσκι. Και τελειώσαμε το σημείο 4. Όπω είπα και στην αρχή, το σημείο 5, η γνωμοδότηση τη κυρίας Μπρίτα Ρέιμερς αναβάλλεται για την συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Και περάμε στο σημείο 6 Σημείο 6, πολύ σημαντικό αγαπητοί συνάδελφοι, ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ε, διαφήμισης σχετικά με τα γεωρικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Θα συζητήσουμε τη νέα πολιτική ενημέρωση και προώθησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για να είμαστε σε θέση ανταγωνιστική με τους εταίρους μας, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, ως εισαγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων, σίγουρα το θέμα της προώθησης θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί εκεί στερούμε. Θα θυμάστε ότι στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα είχαμε ακούσει μία παρουσίαση από τον αρμόδιο επίτροπο τον κύριο Τσόλο και μάλιστα έγινε και μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Γι' αυτό και θα δώσω πάρα αυτό το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Εστέρ Εράνς Γκαρσία. Έχεις το λόγο. Εστέρ και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα που έχουμε περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον περισσότερο από την προηγούμενη Δευτέρα, με τα συγχαρητήρια που θα απευθύνουμε στον Επίτροπο, τον κύριο Τσιόλος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση την οποία καταθέτει και που έχει σκοπό να βελτιώσει τη θέση κάποιων εμπορευμάτων ευρωπαϊκών στις διεθνείς αγορές. Ένας από τους στόχους που είχαμε και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της αιτίας μας. Καλύτερη λοιπόν προώθηση και στην ευρωπαϊκή αγορά των δικών μας προϊόντων μια και οι γεωργοί στην Ευρώπη όλο ένα και περισσότερο αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνισμού με προϊόντα από τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους μέτρα είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος έδειξαν μεγάλη ευαισθησία για αυτή την δύσκολη πραγματικότητα. Άκουσαν και ποιες είναι οι δικές μας διεκδικήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια και εδώ και αρκετό καιρό πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να προετοιμάσουμε αυτή την πρόταση. Αυτές οι εκστρατείες προώθησης ήταν πολύ χρήσιμες ε, για να ξεπεράσουμε την κρίση της ε, βήθησης κάποιων τιμών ή ε, κάποιων υγειονομικών σκανδάλων. Για παράδειγμα, τα όσα συνέβησαν με τα κολοβακτηρίδια ή κόλλη πριν από μερικά χρόνια λόγω κακής συντήρησης προϊόντων μας έδειξαν πως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι για να ξεπεράσουμε καταστάσεις αντίστοιχες με αυτές που ε, βιώσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Το μόνο το οποίο με στενοχωρεί είναι πως δεν είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας γιατί στην ε, ΚΑΠ δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιου είδους εξαρτής προώθηση στο παρελθόν για τα προϊόντα μας. Η πρόταση αυτή βεβαίως και θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά πρέπει να σας πω πως οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι την αντιμετώπισαν πολύ θετικά και η εκτελεστική επιτροπή μοιάζει έτοιμη να προωθήσει τέτοια είδους γεωργικά προϊόντα ε, τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν για εμάς αρκετά σημαντικά και βλέπουμε πως για τις εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Δηλαδή από το 6,1, 61,5 εκατομμύρια ε, τα οποία είχαμε εγγράψει το 2013 στο προϋπολογισμό Φτάσαμε στα 200 κάτι ε, για το 2020, οπότε καταλαβαίνετε πως η αύξηση από τα 61 στα 200 κάτι, 220 είναι ε, ριζική. Επίσης, εμπορικά σήματα, προέλευση, όλα αυτά θα πρέπει ε, να αποτελέσουν ε, στοιχεία ε, υπέρ μας και βεβαίως θα ενταχθούν στην νομοθεσία όπως αυτή εξελίσσεται. Το εμπορικό σήμα, η εμπορική ονομασία και το κράτος προέλευσης είναι μία από τις βασικές διεκδικήσεις του γεωργικού διατροφικού κλάδου, μια και όσο δεν χρησιμοποιούνται δεν μπορούμε να φέρουμε σε πέρα σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε επίπεδο κλαδικό. Θα πρέπει δηλαδή συγκεκριμένε εμπορικέ ονομασίε να προκριθούν και αυτό ενδεχομένω είναι ανησυχητικό για κάποιου. Αν όμω το σκεφτούμε θα δείτε πω τελικά θα ευνοήσει όχι μόνο όσους φέρουν αυτή την εμπορική ονομασία, αλλά συλλογικά όλους τους παραγωγείς ε, του συγκεκριμένου κλάδου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την όθηση που θα δώσουν αυτά τα ονόματα που αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και τρίτες χώρες για να προωθήσουν και τα δικά τους προϊόντα. Θέλουμε λοιπόν μια πιο ανοιχτή και πιο γενναιόδορη πολιτική για, τα, για τις εμπορικές ενομασίες και νομίζω πως η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι ένα μεγάλο ε, βήμα προς τα εμπρός. Ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τι στόχους έχει, δηλαδή πώς θα είναι πιο εμφανής και η προέλευση των προϊόντων αλλά και η εμπορική ονομασία κατά τις εκστρατείες ενημέρωσης και καλό θα ήταν ε, να μας τα πει έτσι ώστε να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι και ο ίδιος ο κλάδος. Θα ήταν αφελές να πιστέψουμε πως οι περιορισμοί της, ε, των κανόνων ανταγωνισμού ε, θα ξεπεραστούν εντελώς με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν αποτελούν την ε, ε, λύση και θα πρέπει την πολιτική ανταγωνισμού να την αντιμετωπίσουμε και από άλλα μονοπάτια, αλλά τουλάχιστον διευκολύνομαστε με κάποια εμπόδια τα οποία μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να υπερπηδηθούν. Τώρα, σχέσεις εμπορικές με τη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, με τον Καναδά, με την ε, Μερκοσούρ, για όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μία σφριγγυλή ευρωπαϊκή ποιότητα ε, θα ήταν ένα στοιχείο πολύ ευνοϊκό ε, για τον κλάδο της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, ε, των διατροφικών προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής ποιες είναι οι ιδιότητες των γεωργικών προϊόντων, των ευρωπαϊκών και με τον τρόπο αυτό να κάνει μια διαφοροποίηση με προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να δώσουμε ευρωπαϊκή προτίμηση, αλλά μπορούμε να ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τη σημασία που έχει ε, να αναγνωρίσει τις προσπάθειες που κάνουν οι δικοί μας γεωργοί και τον αντίκτυπο για την υγεία του και για την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει. Θα πρέπει έτσι να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι προσπάθειες που κάνουν οι επαγγελματίες του κλάδου για να εξασφαλίσουν την ε, ποιότητα των τροφίμων, το περιβάλλον, όπως επίσης και ε, την πτυχή της υγείας. Μία από τις μεγάλες ε, ένα από τα θετικά αυτής της πρότασης είναι αυτή η κεντρική διαχείριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξεπεράσουμε κάποια διαχειριστικά προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν σε εθνικό επίπεδο μεταξύ κρατομελών που δυσκολεύουν αυτού του είδους τις εκστρατείες. Παρ' όλα αυτά, το ότι το 75% των κονδυλίων ε, θα ε, διατεθεί για εξωτερικές δράσεις, νομίζω ότι μειώνει τις προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε στις εσωτερικές αγορές, που είναι η βασική αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όπου οι επαγγελματίες του κλάδου χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μεγάλη, μεγάλο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Αυτό το 75-25 που έχουμε κατανέμει ενδεχομένως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούμε. Συμφωνώ δε πως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι εξωτερικές αγορές αυτή τη στιγμή προσφέρουν τις περισσότερες ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να αναπτυχθούν εκεί τα δικά μας προϊόντα. Αλλά δεν θα πρέπει για το λόγο αυτό να αποστρέψουμε το βλέμμα από την εσωτερική αγορά που σήμερα ουσιαστικά είναι η μεγάλη αγορά για τους δικούς μας παραγωγούς το ότι τα κρασιά έχουν συμπεριληφθεί εδώ, παρόλο που έχουν τα δικά τους κονδύλια τα εθνικά μέσω της κοινή οργάνωσης αγοράς για την ενημέρωση και την προωθήση, ήταν κατά τη γνώμη μου μια πολύ ευφυής ιδέα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω αυτόν τον εμβληματικό κλάδο της γεωργικής παραγωγής Ευρώπη όταν κάνουμε κάποιε δράσεις στο εξωτερικό. Είναι αναγνωρισμένο ο κλάδος παγκόσμια. Η πρόταση βέβαια λέει πως θα έχει δικαίωμα μόνο συμμετοχής σε εκστρατεία, ενημέρωση και προώθησης ε, συνοδεύοντας άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν ο κλάδος αυτός θα είναι ο μοναδικός ευρωπαίος παραγωγός που δεν θα μπορεί να κάνει αποκλειστικά εινοπαραγωγικές εκστρατείες ε, σε προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν περισσότερο από ένα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θα μπορούσε να το ξαναδεί γιατί ο κλάδος έχει ήδη καταγγείλει ε, το γεγονός αυτό γιατί στις ε, εκστρατείες που κάνουν πολλές χώρες μαζί είναι πολύ μικρό το μερίδιο το οποίο έχει διατεθεί για ε, τα κρασιά γιατί οι χώρες σε αυτό τον κλάδο δεν συντονίζονται μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική ευρωπαϊκή που θα λύνει το πρόβλημα αυτό και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες σκέψεις να μοιραστεί μαζί μας. Επίσης δεν επιτρέπεται πλέον η εθνική συγχρηματοδότηση των μέτρων πρόθεσης και ενημέρωσης και αυτό δημιουργεί ανησυχίες. Ο παραγωγικός κλάδος φοβάται πως θα χρειαστεί να συνεισφέρει περισσότερο ο ίδιος. Ρωτώ λοιπόν τους συναδέλφους ποια είναι η άποψή τους και ρωτώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν ανησυχεί μήπως ένα μέτρο τέτοιου είδους θα ευνοήσει περισσότερο τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ε, περισσότερους πόρους στις, ε, στη διάθεσή τους, δηλαδή αυτούς με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Μήπως θα έπρεπε να αυξήσουμε τη συγχρηματοδότηση για τα μέτρα προώθησης, για παράδειγμα όταν έχουμε γεωργικές κρίσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε συνθήκες διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών ε, που έχουν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και αυτών που έχουν πιο περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους. Να μας ξεκαθαρίσει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος είναι ο στόχος της. Πώς θα έχουμε καλύτερη και ταχύτερη αντίδραση και πιο ευέλικτη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τέτοιων ε, προβλημάτων και κρίσεων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε πως δεν έχει εργαλεία και δεν έχει ταχεία αποτελεσματική και αποδοτική αντίδραση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά. Η πρόταση διευρύνει το πρώτο παράρτημα του, ε, της συνθήκης με τον κατάλογο προϊόντων που μπορούν να συμπεριληφθούν στις εκστρατείες προώθησης και κάποια μεταποιημένα τα οποία είναι πλέον επιλέξιμα ε, στα πλαίσια των ε, καθεστώτων ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν θα ήθελα να μου πούν οι συνάδελφοι τι πιστεύουν. Είναι ε, απαραίτητο το παράρτημα να διευρυνθεί, δηλαδή να αυξηθούν τα προϊόντα που είναι στον κατάλογο του ε, παραρτήματος για την ε, Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή που θα διαχειρίζεται αυτές τις δράσεις. Δεν είμαι κατά, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να στήσουμε ένα καινούριο φορέα εδώ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους, να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες που έχουν ήδη στηθεί και με τον τρόπο αυτό να βρούμε συνέργειες με τα στοιχεία και τα εργαλεία τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας ε, διευκρινίσει ποια θα είναι η πρικοδότηση του μέτρου και πώς θα χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, θα καλύψουμε και τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα της διαχείρισης μέσω των κονδυλίων για την προώθηση το να τρέχει κεντρικά το πρόγραμμα επιλογής ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικό. Γιατί μιλάμε για εκστρατείες που θα διαχειρίζεται και θα τρέχει ένα κράτος μέλος. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ένα βήμα πίσω και αφού ε, θα κάνει την ίδια την εκστρατεία προώθηση και θα το διαχειρίσει, να αφήσει τα κράτη-μέλη την επιλογή. Και τέλο, θέλω να σα πω πω η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εργασία ετήσιο μα βρίσκει σύμφωνος γιατί έτσι θα έχει μια σαφή στρατηγική αυτή η πολιτική πρόθεση, κάτι που έλειπε μέχρι σήμερα και νομίζω ότι καλό είναι να συγχαρούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αποφάσισε να έχει και να δημιουργήσει και μια πλατφόρμα καθοδήγησης ε, του κλάδου ε, και να δημιουργήσει και ένα σλόγγαν ευρωπαϊκό για καθένα προϊόν. Νομίζω ότι για τα λογότυπα και για τα αναγράμματα και για τα σλόγγαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάνει πολλή δουλειά και θα πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας χρησιμοποιώντας ό,τι ήδη υπάρχει χωρίς να δημιουργήσουμε ε, παραπάνω πληροφορίες τις οποίες θα ε, δυσκολευτούμε να περάσουμε ε, στον καταναλωτή. Επαναλαμβάνω, την πρόταση αυτή θα τη δεχτούμε πολύ θετικά. Είναι καλή η πρόταση και βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί με τη συνεισφορά τη δική μας μέσω των σχολείων των συνοδέλφων και με μεγάλη χαρά περιμένω τα δικά σας σχόλια, συνάδελφοι. Ε, Ωραία, ευχαριστούμε κυρία Ρας έχουν ζητήσει το λόγο μερικοί συνάδελφοι. Περνάμε στη συζήτηση. Πρώτος ο Τζιμ Νίκολσον. Έχεις το λόγο, Τζιμ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεση και την uh, αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού στον τομέα, πράγμα όλος ευπρόσδεκτο. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εξωτερική και όχι στην εσωτερική πρόθεση γιατί εκεί υπάρχει θετική μεγέθυνση και από εκεί θα προέλθει η απόδοση των επενδύσεων μακροπρόθεσμα. Άλλωστε είναι ο τομέας όπου πρέπει να επικεντρωθούμε αφού οι διεθνείς αγορές δεν πρέπει να πάνε σε χέρια άλλων. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τα αγαθά που παράγουμε στην Ευρώπη. Για τη συγχρηματοδότηση, σίγουρα καλωσορίζω το τέλος της, γιατί ε, ήταν μια υπερβολική υπεραπλούστευση ε, χρησιμοποίηση πρόσθετων κονδυλίων από την περιοχή ε, υπήρχε. Νομίζω λοιπόν ότι θα περιορίσουμε τους μεσάζοντες έτσι και θα έχουμε πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό μακροπρόθεσμα. Οι μικροί παραγωγοί θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στους μικρούς παραγωγούς που θα έχουν πρόσβαση και οι μικροί συνεταιρισμοί θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα και θα γίνεται καλή προώθηση από εθνικούς διάβλους σε επίπεδο κράτους μέλους και θα έχουν την ευκαιρία να ε, έχουν πρόσβαση σε, αυτό το, σε αυτή τη χρηματοδότηση. Δεν θα υπάρχουν οργανισμοί για να ε, διευκολύνουν αυτό το ταμείο. Αυτό είναι καλό γιατί έχουμε υπερβολικούς οργανισμούς και δεν χρειάζονται άλλοι. Ε, Είμαι λοιπόν υπέρ αυτής της θέσης που έλαβε ο Επίτροπος. Επίσης είμαι υπέρ της κίνησης να συμπεριληφθούν μεταποιημένα προϊόντα στον κατάλογο. Σημαντικό αυτό ιδιαίτερα για τους τοπικούς παραγωγούς. Θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα τη θέση τους. Προσοχή όμως ε, μην ε, το παρακάνουμε με τη χρηματοδότηση, τα κονδύλια θα γίνουν έτσι αναποτελεσματικά. Είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός πάντοτε όταν πρόκειται για νέα προγράμματα, νέες ε, ε, δράσεις. Δηλαδή θα γίνει τόσο ισχνή διασπορά των κονδυλίων που γίνεται αναποτελεσματική. Πρέπει να είναι πιο στοχευμένες οι πιστώσεις μας, τα κονδύλια που παρέχουμε. για να είναι αποτελεσματικά. Επίσης, ε, υπάρχουν και άλλα θέματα ε, το Made in Europe ε, γίνεται πολύ λόγος γι' αυτό. Τι σημαίνει, πρέπει να αναρωτηθούμε. Ε, σίγουρα έχει νόημα αυτό για κάποιες επωνυμίες. Να προωθηθεί δηλαδή το ευρωπαϊκό προϊόν. Αλλά μέσα στα κράτη-μέλη, στις εγχώριες αγορές, σίγουρα αυτό θα υπονομεύσει τα ντόπια προϊόντα και αν δείτε τη μεγάλη ε, διαφορετικότητα σε όλη την Ευρώπη, τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων από, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, είναι σημαντικό αυτή η ποικιλομορφία να μην αλλάξει ε, μέσα από ε, οριζόντιες επωνυμίες ευρωπαϊκές. Επίσης υπάρχουν κάποιες ε, μοναδικές επωνυμίες, ε, τα Ιταλικά, τυριά, το κρέας στη Σκοτία, βόλιο κρέας, ε, νομίζω ότι αυτά είναι προϊόντα αναγνωρισμένα από πολλά χρόνια και δεκαετίες. Η πρόταση θα πρέπει να προωθεί τα προϊόντα στις αγορές χωρίς να παραγνωρίζει την εξαιρετική δουλειά που έγινε για την ανάδειξη μεμονωμένων επωνυμιών υψηλής ποιότητας. Ε, αυτό ε, είναι σημαντικό να μην ανατραπεί. Αυτή είναι η θέση μου, κύριε Πρόεδρε. Θα χαρώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και θα υποβάλω ένα ε, πρόγραμμα σχέδιο προτάσεων που θα ε, αυξήσουν το μέγεθος ε, της αγοράς για τα προϊόντα που παράγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ράς Γκαρσία Περές. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια με κάλυψε με τα όσα είπε γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά θέματα που προκύπτουν από την έκθεση δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θέλω να την ευχαριστήσω για την τόσο λεπτομερή της ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι συμπίπτουμε όλοι στην άποψη πως ο κανονισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός και ο στόχος που έχουμε για την προώθηση των προϊόντων της Ευρώπης, των γεωργικών προϊόντων, είναι σε μία πρώτη φάση να κλείσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την ποιοτική διάσταση των προϊόντων. Αυτό είχε μείνει, ε, εάν θέλετε, ανοιχτό ε, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για την ΚΑΠ. Άρα λοιπόν τα θέματα αυτά είναι ουσιαστικά, αντιμετωπίζονται πολύ σωστά, είναι η εμπορική ενομασία και η προέλευση που θα πρέπει να στηρίξουν αυτές τις εκστρατείες, οι ενώσεις παραγωγών που αναλαμβάνουν ρόλο, και για την διαβούλευση στην οποία αναφέρθηκε η συγγήτρια για τα όσα είπε καταρχήν για τον εινοπαραγωγικό κλάδο, συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κλάδο αυτό ε, με διακρίσεις. Θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στην προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων όπως οι υπόλοιποι ένα θέμα στο οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι η δυνατότητα ή όχι της συγχρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείει αυτή την δυνατότητα και θεωρεί πως θα ήταν πολύ πιο ευέλικτο ε, και πολύ πιο απλό στη διαχείριση αν δεν έχουμε έλεγχο από πλευράς ε, κρατών μελών, αλλά εξακολουθώ να αμφιβάλλω το κατά πόσο χρειάζεται ή όχι δεν είμαι σίγουρη. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις καλό είναι τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στα, στις προσπάθειες αυτές προώθησης. Κάτι το οποίο δεν μου έχει γίνει ακόμα σαφές και ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να αποκλείσουμε εξ αρχής είναι η δυνατότητα συμμετοχής έτσι ώστε να καλύψουμε ένα διπλό στόχο, δηλαδή και την απλούστευση της διαχείρισης αυτών των σχεδίων, αλλά παράλληλα και την δυνατότητα που θα ανοίξουμε στα κράτη-μέλη συμμετοχής σε αυτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος γιατί οι εισηγήτρια και οι προλαλήσαντες με κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό. Δύο θέματα θα θέσω. Είναι νομίζω σωστό στο βαθμό του δυνατού και όσο γίνεται περισσότερο τα διαθέσιμα χρήματα να τα δώσουμε στους επιχειρηματίες στην αγορά. Δεν πρέπει οι Βρυξέλλες να κάνουν διαφημιστικές εκστρατείες για προϊόντα που υπάρχουν στις εγχώριες αγορές. Ε, γιατί δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή αγορά για μπανάνες ή για μήλα ή για κρασί. Υπάρχουν κάποιες ορατές μάρκες για τους καταναλωτές και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσουμε αποτελεσματικά ε, τα προϊόντα, τα προϊόντα στον καταναλωτή και όταν πηγαίνει ο τελευταίος στο ε, σούπερ μάρκετ να τα βλέπει εκεί. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό με τα ευρωπαϊκά κονδύλια να ε, προωθήσουμε τις μάρκες που είναι δικές μας. Ε, δηλαδή αυτές που υπάρχουν στην δέσμη ποιότητας και αποφασίστηκαν είναι οι ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις, τα βιολογικά, ε, είναι οι ευρωπαϊκές ονομασίες, είναι το δημόσιο αγαθό ιδιοκτησία μας, η περιουσία μας και είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προωθήσει στην αγορά τις επωνυμίες αυτές. Οι υπόλοιπε θα πρέπει να προωθούνται από τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε με το εγχείρημα προώθησης ποιοτικών προϊόντων στην αγορά. Ευχαριστώ. Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για Ευρώπη και ευρωπαϊκά, είναι αμφιλεγόμενος όρος όταν προωθούμε προϊόντα. Μπορεί να είναι και ανακριβής. Υπάρχουν 8-9 χώρες στην Ευρώπη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έλεγα τα οι Βρετανοί φορολογούμενοι να προωθούν προϊόντα από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 4 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι στην Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα εδώ. Οπότε η λέξη Ευρώπη-Ευρωπαϊκός ε, είναι λέξεις που πρέπει να εξεταστούν κάπως πιο προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τον κύριο Φερστέιλεν. Α, συγγνώμη, ζήτησε το λόγο πρώτα ο κύριος Καπόλας Άντος και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Άγνιο που είπε ότι δεν συμφωνεί τα χρήματα των φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου να χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε όμως κύριε Άγνιου τα χρήματα των φορολογουμένων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν βρετανικά προϊόντα. Αυτό δεν σας ενοχλεί. I would Πολύ ευχαρίστω ε, αν ε, ε, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Έλληνες, Γάλλοι συσπηρωθούν και προωθήσουν βρετανικά προϊόντα. Αλλά δεν λειτουργεί το σύστημα. Η Μεγάλη Βρετανία συνεισφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να βοηθήσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο διευθυντή ο κ. Βερστάιλεν και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Ράζ Καρσία, την εισηγήτριά μας. Παρακαλώ κύριε Βερστάιλεν. Okay. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και αρχίζω... Να ξεκινήσω με το θέμα της χρηματοδότησης. Γιατί προτείνεται η κατάργηση της χρηματοδότησης. Κυρίως η χρηματοδότηση για το τμήμα της συνεισφοράς των κρατών μελών. Αυτή η χρηματοδότηση συνιστούσε εξαίρεση στο γενικό κανόνα από τα μέτρα του πρώτου πυλώνα. Και θελήσαμε να καταργήσουμε αυτή την εξαίρεση. Επίσης, είναι συνέπεια μιας προσπάθειας απλούστευσης που κάνουμε για την επιλογή των προγραμμάτων, που γίνεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να περνάμε από τα κράτη-μέλη. Στο προηγούμενο, το παλιό σύστημα, η δημόσια χρηματοδότηση μπορούσε να φτάσει μέχρι το 80%. 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 30% από τα κράτη-μέλη. Ε, μερικές φορές όμως είχαμε ελάχιστη ε, ανάληψη ευθύνης από τους προτείνοντες και λίγα προγράμματα. Οι εθνικές άλλωστε συγχρηματοδοτήσεις είχαν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεχίσουν παρόλα αυτά να χρηματοδοτούν τα προγράμματα, τα δικά του προγράμματα πρόθεση των γεωργικών του προϊόντων, φυσικά με σεβασμό των ε, ισχυών των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσει. Άλλο θέμα σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό της εσωτερικής αγοράς από την αγορά των τρίτων χωρών και γιατί δίνουμε έμφαση στις ε, δράσεις της ε, τρίτες χώρες. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Για τις εξωτερικές αγορές έχουμε, ε, δίνουμε προτεραιότητα για να βρούμε νέες διεξόδους, προασπίζοντας τον επιστηστικό μας κλάδο και αναπτύσσοντας την ανταγωνιστική του θέση στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και οι δράσεις στις τρίτες χώρες προωθούνται, αλλά είναι πιο δαπανηρές. Δεν ξεχνούμε φυσικά την εσωτερική αγορά και θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του Ευρωπαίου καταναλωτή. Να προσθέσω επίσης ότι σήμερα δαπανούμε μόνο το 30% το κονδυλίων για τις τρίτες χώρες. Ε, κατά τη γνώμη μας είναι πολύ ισχνό αυτό το ποσοστό. Άλλωστε, στα πλαίσια της ε, εξωτερικής αγοράς δεν χρησιμοποιούμε πια το μηχανισμό των εξαγωγικών επιστροφών. Έχουν σχεδόν καταργηθεί εξαγωγικές επιστροφές. Επίσης, ε, οι περισσότερες ε, δυνατότητες ανάπτυξης βρίσκονται στις τρίτες χώρες. Μέχρι το 2050, η, αύξηση των γεωρικών μας ε, εισαγωγών, εξαγωγών προς χώρες ΑΣΑΝ θα ήταν μέχρι και 17 δισεκατομμύρια το χρόνο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρτί που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ για την πολιτική αυτή και σε καμία περίπτωση δεν θα βρεθεί χαμένη μια αγορά. Παντού θα αυξηθεί η προώθηση και μάλιστα με ένα προπολογισμό 200 εκατομμύρια μέχρι και 25% δηλαδή 50 ε, εκατομμύρια θα έχουμε για την εσωτερική αγορά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι αφιερώνουμε σήμερα για τα μέτρα της εσωτερικής αγοράς. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν παραμελούμε ή δεν ξεχνούμε την εσωτερική αγορά. Αλλά διαπιστώσαμε ότι όταν γίνεται η προώθηση ενός προϊόντος στην εσωτερική αγορά εκτοπίζεται αυτόματα άλλο προϊόν. Ενώ στις εξωτερικές αγορές, στις αγορές των τρίτο χωρών δηλαδή, αναζητούμε νέες διεξόδους. Οπότε αυξάνονται οι δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπορικό σήμα και το θέμα της προέλευσης και πώς τα εμπορικά σήματα θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκστρατεία της προώθησης. Στα πλαίσια του οριζόντιου καθεστώτος προώθησης, η συγχρηματοδότηση προτιμά, απαιτεί ένα γενικό ευρωπαϊκό μήνυμα, γιατί το δικό μας σύστημα προώθησης συμπληρώνει ουσιαστικά τα υπόλοιπα προγράμματα προώθησης. Και θέλουμε να στείλουμε ένα ευρωπαϊκό μήνυμα που συμπληρώνει τα υπόλοιπα μηνύματα. Βέβαια τα εμπορικά σήματα μπορούν να παραμένουν ορατά, υπό τον όρο όμως ότι έχουμε περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα και ε, το ένα δίπλα στο άλλο, όχι ένα βασικό μήνυμα. Το βασικό μήνυμα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό, αλλά μπορούν να είναι εμφανίσιμα και τα υπόλοιπα ορατά και τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα. Γιατί πολύ συχνά τα προϊόντα μας φέρουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Πάντως η πρόθεση αυτή των προϊόντων μας δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση τη χρήση μόνο εμπορικών σημάτων. Θα πρέπει πάντα να συνοδεύονται αυτά με το ευρωπαϊκό μήνυμα κατά κάποιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την προέλευση τώρα. Θεωρούμε ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να τηρηθούν και έχουμε και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα της προέλευσης. Για τα προϊόντα με γεωγραφική συγκεκριμένη προέλευση, μία αναφορά της προέλευσης μπορεί να γίνει όπως προβλέπεται στον γεωργικό εντοπισμό. Επιτρέπεται μία τέτοια αναφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, η προέλευση θα πρέπει να αναφέρεται ως δευτερεύον μήνυμα σε σχέση με το γενικό ευρωπαϊκό σήμα. Και για τις τρίτες χώρες η προέλευση μπορεί να αναφέρεται στο βασικό μήνυμα, αλλά μαζί με το γενικό ευρωπαϊκό μήνυμα, στο ίδιο επίπεδο δηλαδή. Οπότε θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να προβάλλουμε αυτή την ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με κάθε τρόπο. Επιλογή των προγραμμάτων ποια είναι η ισχύουσα διαδικασία για την επιλογή των προγραμμάτων. Όπως θα διαπιστώσετε και από την πρότασή μας, στόχος μας είναι η απλούστευση. Δηλαδή θέλουμε μια διαδικασία με μονοπευθυντική θηρίδα, δηλαδή με επιλογή των προγραμμάτων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε την ε, ισχύουσα διαδικασία με τα δύο στάδια, πρώτα τα κράτη-μέλη και μετά η Επιτροπή και θέλουμε μία φορά το χρόνο και όχι δύο φορές το χρόνο, δύο φάσεις μέσα στο χρόνο. Με το πρόγραμμα έχουμε μεγαλύτερη απλούστευση, κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη, μετά όμως την προεπιλογή που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έχουμε μία ενιαία δίωδο προεπιλογής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά τα πολλαπλά προγράμματα, προτείνουμε άμεση διαχείρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί προτείνουμε τώρα να απομακρύνουμε τα κράτη-μέλη από την προεπιλογή των προγραμμάτων. Γιατί οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και δαπανηρές για τους δικαιούχους. Θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες των δικαιούχων, προσφέροντας μια διαδικασία επιλογής ε, πολύ πιο ταχεία. Διαπιστώσαμε μάλιστα από την εμπειρία μας ότι η διαδικασία με τις δύο φάσεις ε, έχει όρια. Και μερικές φορές είναι ανεπίτρεπτη η επικάλυψη που γίνεται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της άμεσης διαχείρισης των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουμε και τη χρήση ενός ε, ε, εκτελεστικού γραφείου. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια, ένα νέο οργανισμό ε, για τα εκτελεστικά αυτά καθήκοντα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες οργανισμούς. Έτσι θα αυξηθεί η ικανότητά μας για άμεση διαχείριση για τα προγράμματα αυτά και για την τεχνική υποστήριξη, γιατί ε, υπάρχουν πολύ πιο ειδικευμένοι φορείς για την ε, εκτέλεση εκστρατιών ε, πρόθεσης. Ε, άνθρωποι πολύ πιο ειδήμονες για το θέμα αυτό από ότι πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τη στιγμή που αυξάνονται οι δαπάνες, προτείνουμε τα 200 εκατομμύρια, θα χρειαστούμε και περισσότερο προσωπικό για την διεξαγωγή αυτής της πολιτικής πρόθεσης. Προκειμένου λοιπόν να εξορθολογήσουμε την πολιτική και μετά από μια ανάλυση κόστους ωφέλους, προτείναμε εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης σε έναν εκτελεστικό οργανισμό. Έτσι θα κάνουμε και κάποιες οικονομίες σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Επίσης ε, θα εμπλουτίσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στα θέματα πρόθεσης των προϊόντων. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εφαρμόσει μια ταχύτερη διαδικασία επιλογής και μάλιστα και εσείς ε, ζητήσατε έχουμε άμεση ανταπόκριση με την καλύτερη δυνατή διαδικασία. Πιστεύω ότι η προτινόμενη διαδικασία είναι η καλύτερη και η ταχύτερη. Γιατί μεσούς της κρίσης ε, λαμβάνουμε μερικές φορές και έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και εδώ εμπίπτει και η πρόθεση είχαμε ε, περιπτώσεις όπως τη, την επιζωτία στα πουλερικά ή και τα κολοβακτηρίδια, τα εσχερίδια κόλλη. Εκεί χρειάστηκαν κάποια μέτρα, αλλά επειδή ακριβώς έπρεπε να περάσουν αυτά από τα κράτη-μέλη, πέρασε πολύ σκερός μέχρι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα πρόθεσης. Ήδη έχουμε ξεπεράσει την κρίση πριν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα με τόσο χρονοβόρες διαδικασίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα μας πρόταση για μόνο απευθυντική θηρίδα θα μπορέσουμε να τη δούμε πιο άμεσα και πιο γρήγορα ακόμη και σε περίπτωση κρίσης. Τέλος, δύο λόγια για τη, χρηματοδότηση, για τη συγχρηματοδότηση. Επαναλαμβάνω, προτείναμε κατάργηση της συγχρηματοδότησης για να επιταχύνουμε τη διαδικασία επιλογής κυρίως. Γιατί τώρα η Επιτροπή θα αποφασίζει απευθείας για τα διάφορα προγράμματα πρόθεσης. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να απαιτούμε συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν λόγο σε αυτήν την επιλογή. Και φυσικά εδώ θα ζητήσουμε άμεσα από τους δικαιούχους να συμμετέχουν κατά 50% οπότε θα αναλαμβάνετε πολύ πιο μεγάλη ευθύνη από αυτούς. Ενώ στο παρελθόν 80% της συγχρηματοδότησης προερχόταν από δημόσιες ενισχύσεις. Στο μέλλον θα έχουμε μόνο 50% δημόσια ενίσχυση και το υπόλοιπο 50% θα το χορηγούν οι δικαιούχοι. Έτσι αυξάνεται και το δικό τους επίπεδο ευθύνης. Ένα τρίτο στοιχείο επίσης σημαντικό στο πλαίσιο αυτό είναι ότι είχαμε κάποιες χώρες που χρησιμοποιούσαν κρατικές ενισχύσεις για το θέμα αυτό. Άλλες χώρες δεν το έκαναν Οπότε ουσιαστικά δημιουργούνταν μια διακριτική μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων εμπόρων ανάλογα με το κράτος προέλευσής τους. Θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια στρέβλωση. Στο μέλλον θέλουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και ίση μεταχείριση για όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ράσκανσία, για τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Δεν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που σας κάναμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σας ευχαριστώ πάντως για τις ε, διευκρινήσεις που μας δώσατε. Ε, ε, από τα όσα απαντήσατε για την συγχρηματοδότηση, νομίζω εδώ θα γίνει πολλή συζήτηση, το είπε και η κυρία Γκαρσία Πέρες, είναι ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε πιο πολύ. Σε κάτι έχετε δίκιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν οι φορείς συνεισφέρουν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι πιο υπεύθυνοι και θα έχουν και πολύ μεγαλύτερο συμφέρον από το να προωθήσουν τα προϊόντα τους εφόσον έχουν επενδύσει ε, μεγάλα ποσά. Αυτό το οποίο δεν ε, με επίθει είναι το κατά πόσο το να αποκλίνουμε τα κράτη-μέλη από τη χρηματοδότηση είναι καλό ε, στο επίπεδο επιλογής των προϊόντων, γιατί εάν χρειάζεται να κάνουν τον έλεγχο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ποια έχουν επιλογή εν πάση περιπτώσει θα συζητήσουμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες το θέμα έτσι ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατόν συνένεση και εν ώψη, του εγγράφου το οποίο θα καταθέσω αργότερα για το 75-25 και την κατανομή αυτή εξακολουθώ να πιστεύω πως από το 30% που δίνεται για την προώθηση σε τρίτες χώρες να πάμε στο 75% η ψαλίδα είναι μεγάλη και νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλύτερη διαπραγμάτευση για το πώς θα μοιραστούν τα κονδύλα, γιατί σας άκουσα, αλλά και η εσωτερική προώθηση, όπως είπε ο συνάδελφος, είναι σημαντική. Η ενημέρωση δηλαδή της ευρωπαϊκής αγοράς. Νομίζω λοιπόν πως θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε αυτά ε, σε επίπεδο Επιτροπής Γεωργίας για να δούμε τι ποσοστό θεωρούμε πως θα έπρεπε να διαθέσουμε για την προώθηση σε τρίτες χώρες και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πω πως οι τρίτες χώρες είναι πολύ πιο δαπανηρή η προώθηση. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι το θέμα αυτό καλό είναι να το ξανασκεφτούμε. Ο κύριος Διευθυντής όταν μιλάει για απλούστευση έχει δίκιο. Είναι πραγματικά ο πρωταρχικός μας στόχος και σχεδόν με έπεισε πως με μία πρόσκληση μόνο ετήσια θα είμαστε πιο ευέλικτοι γιατί θα έχουμε λιγότερες γραφειοκρατικές ε, περιπέτειες αντίθετα με το κάθε έξι μήνες που έχουμε τώρα, αλλά αυτή η σημαντική θηρίδα ε, μου φαίνεται ότι είναι κάπως ρηψοκίνδυνη. Ε, εν πάση δεν θα αποτελέσει και κάουσος μπέλη μεταξύ μας για την εκτελεστική επιτροπή, το είπε και ο κ. Νίκολσον, μας το εξήγησε και ο Επίτροπος την περασμένη εβδομάδα και συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον. Δεν χρειάζεται εμείς να στήσουμε νέες υπηρεσίες, δεν χρειαζόμαστε περισσότερη γραφειοκρατία. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε και δεν χρειάζεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει τα χρήματα να χρησιμεύσουν στους πολίτες, από όπου και να προέρχονται στους Ευρωπαίους πολίτες με λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη ε, διαχείριση. Για το πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις δεν το είπε πολύ ανοιχτά ο κύριος Διευθυντής, αλλά η κατεξιοδότηση πράξη κατά τη γνώμη σας αποτελούν τη λύση για ταχεία αντίδραση. Εμένα δεν με ικανοποιούν πολύ αυτές οι κατεξουσιοδότηση οι αναθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρουν συνάδελφοι πως πάντα αντιδρώ. Αλλά εάν τουλάχιστον με τον τρόπο αυτό καταφέρουμε ο κλάδος αυτός να μην πλήττεται όπως σήμερα από την γραφειοκρατία μεταξύ κρατών μελών, τότε έχει καλός. Ίσως όμως μπορέσουμε να εφεύρουμε και κάποιο άλλο σύστημα που θα μπορούσε να ξεπεράσει τους περιορισμούς των κατοξουσιοδότηση πράξεων. Η κυρία Ιράτσα Γκαρσία έχει δίκιο. Μας έλειπε όντως η διάσταση της ποιότητας ε, και μην ξεχνάτε τα όσα έχουμε στο πακέτο ποιότητας όπου ο στόχος είναι η απλούστευση του συστήματος για τα εμπορικά σήματα, για τα εμβλήματα, για τα λογότυπα που χρησιμοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε καινούρια, να βρούμε τις ενέργειες μεταξύ τους έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο και προσπάθειες, γιατί στο κάτω-κάτω θα κατανοίξουμε σε νέα λογότυπα τα οποία δεν θα αναγνωρίζει κανείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξορθολογήσουμε ε, την ε, δράση μας και να μην φτιάξουμε καινούρια σχεδιάκια τα οποία θα κολλάμε ε, πάνω στις σημάνσεις για τη μη διακριτική μεταχείριση του υνοπαραγωγικού κλάδου έχετε δίκιο. Είναι μια διάκριση και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει. Θα ήθελα να ε, διασκεδάσω τις ανησυχίες του κυρίου Άγνιου είναι για τα ευρωπαϊκό προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Τώρα η Ουκρανία και η Λευκορωσία είναι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, άρα λοιπόν εμείς θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε όσους βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα τα κράτη-μέλη έχουν αρκετά το αριθμό προϊόντων, είτε κτηνοτροφικά, είτε γεωργικά, είτε διατροφικά, για να δρέψουν τα πλεονεκτήματα αυτού του πακέτου. Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο στόχος της εισηγήτριας και πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα με συνοδεύσει σε αυτή την προσπάθεια να γίνουν πιο αναγνωρίσιμοι ε, τα αναγνωρίσουμε τα προϊόντα αυτά και να αναγνωρίζεται και η ποιότητά τους. Θα κάνουμε τις συνεδριάσεις με όλους τους ε, σκιώδες εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες και βεβαίως και με τους βουλευτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έκθεσή μου ακόμα και αν δεν είναι σκιώδες εισηγητές, γιατί είναι σημαντικό τις ιδέες όλων να τις συλλέξουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατόν συνένεση και να έχουμε τον ελάχιστο αριθμό τροπολογιών. Το πακέτο αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και ίσως μπορεί να μας δώσει και σε μια ευκαιρία να το ε, βοηθήσουμε να προχωρήσει. Δεν θέλουμε ένα τεράστιο φάκελο με πολλές τροπολογίες. Θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Σας ευχαριστώ. Και στόχος μας είναι το θέμα να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση το συντομότερο δυνατόν και επαναλαμβάνω με τη μέγιστη δυνατόν συνένεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ραντ Καρσία. Ευχαριστώ και του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο σημείο 7 τη της διάταξη αλλά δεν έχει έρθει ακόμη ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα κάνουμε μια δεκάλεπτη διακοπή και μετά θα ακούσουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, ένα δεκάλεπτο διάλειμμα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

Κούφετ. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης ε, είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2013. Η νέα στρατηγική θα επικαιροποιήσει και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα στρατηγική τα δάση του 1998 με γενικότερο στόχο της ε, ανακοίνωσης ε, η κατάρτιση μιας στρατηγικής ε, για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα στηρίζεται στη έννοια της αϊφόρου διαχείρισης των δασών και στον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον ε, κύριο Χόλτσερ από τη Γενική Διεύθυνση, με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, τμήματάρχη του Τμήματος Βιοεργίας, Βιομάζας, Δασών και Κλιματικών Αλλαγών, που θα μας παρουσιάσει τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Κύριε Χόλτσερ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου επίσης. Καταρχήν, Εκφράζω ευγνωμοσύνη διότι προλάβαμε και φέτος να έρθουμε και να παρουσιάσουμε τη δασική στρατηγική, ένα έργο που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια με εντατικού ρυθμούς και ολοκληρώθηκε, όπως είπατε, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, με την έγκρισή του από την Κομισιόν στις ε, 20 Σεπτεμβρίου. Θα παρουσιάσω το περιεχόμενο εν συντομία και κάποια επόμενα βήματα που προβλέπουμε. Η δασική στρατηγική, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι καινούρια. Άρχισε το 98 να υπάρχει και τώρα αναθεωρείται. Γιατί, Γιατί ο κόσμος άλλαξε σε ό,τι αφορά δασοκομεία και δάση και αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η σημασία των δασών. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, θεωρήσαμε ότι η δασική στρατηγική ως έχει ή ως είχε, ε, είχε εν πολλής ξεπεραστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, και αυτό είναι σημαντικό, ε, τονίζει ότι έξι επιτροποί στηρίζουν την νέα πρωτοβουλία και στρατηγική. Δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται στη δασική κοινότητα μόνο, αλλά έχουμε και την DG Agri καθήλυνα αρμόδια, αλλά και δύο ακόμη ε, συναρμόδιες γενικές διευθύνσεις για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον και η Γενική Διεύθυνση Κλίμα, Ενέργεια και RTD. Αυτό από την αρχή ήταν η πιο σημαντική μας επιδίωξη. Να μην έχουμε δηλαδή μονοπρισματική θεώρηση, αλλά να δούμε όλες τις απόψεις που θα συμβάλλουν στην διάρθρωση της νέας δασικής πολιτικής. Τώρα υπάρχει ένα κείμενο που συνοδεύεται από δύο έγγραφα εργασίας υπηρεσιακά. Το ένα που συνοδεύει την ανακοίνωση για τη νέα βασική στρατηγική και ένα έγγραφο εργασίας υπηρεσιακό για ένα σχέδιο ε, των βιομηχανιών που εξαρτώνται από τη δασοκομεία. Τώρα για το περιεχόμενο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η προσέγγιση που επιλέξαμε. Μιλάμε για δασική στρατηγική, για τα δάση και τον τομέα της δασοκομείας και αυτό που στηρίζεται στα δάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης πολύ σημαντικό είναι η ολιστική προσέγγιση που έχουμε στα δάση και όλων των πολιτικών που αφορούν τη, τα δάση και που περιλαμβάνει και την αξιακή αλυσίδα. Όταν μιλάμε για ολιστική προσέγγιση, τι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και συμπεριληφθεί τελικά. Στο επίκεντρο τα δάση και οι δραστηριότητες ε, περί τα δάση, αλλά υπάρχει και ένας κλάδος ε, δασικής έρευνας και καινοτομίας. Έχουμε το, τα δάση και το περιβάλλον, έχουμε τις βιομηχανίες που στηρίζονται στα δάση, δάση και βιοενέργεια, δάση και αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη υπαίθρου και τέλος δάση και κλιματική αλλαγή και γι' αυτό είναι έξι οι επίτροποι που στηρίζουν αυτή τη δασική στρατηγική. Τώρα, πολύ σύντομα, αυτή η στρατηγική τι θέση έχει και τι στόχους περιλαμβάνει. Καταρχήν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δάση θα παίξουν θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ανάπτυξη, απασχόληση, προστιθέμενη αξία, οικοσυστημικές υπηρεσίες. Πρέπει επίσης να ε, ακολουθήσουμε και τη βασική ενωσιακή πολιτική, στρατηγική πολιτικής, και στην ε, στρατηγική 2020 έχουμε και άλλους στόχους για το 2020 και για το 2050. Έχουμε λοιπόν ε, καλή θεμελίωση στις στρατηγικές μας αυτών των ε, ενωσιακών πολιτικών στόχων. Επίσης, Ε, αυτή είναι ευρωπαϊκή πολιτική που αντικατοπτρίζει και επηρεάζει, όπως ελπίζομαι, όσα λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη, γιατί η δασοκομεία, όπως γνωρίζετε, είναι αρμοδιότητες κρατών μελών, αλλά και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Και κάναμε μακρές συζητήσεις για την επικουρικότητα, βέβαια, όπως και άλλα σημαντικά θέματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η στρατηγική πρέπει να εκλαμβάνεται ως κρίκος σύνδεση ε, των ε, υπολείπων πολιτικών μας και θέλουμε η στρατηγική αυτή να επηρεάσει τη δράση μας για τα δάση σε τομείς ευρωπαϊκής αρμοδιότητας βέβαια, ούτω ώστε να αποστέλλονται τα σωστά μηνύματα. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές αρχές. Πολύ σύντομα θα αναφέρω τρεις βασικές. Πρώτον, η αηφόρος διαχείριση των δασών, δεύτερον αποτελεσματικότητα των πόρων και τέλος η ε, συνολική ε, ευθύνη για τα δάση. Θα δεν θα επισέλθω στις τρεις αρχές τόσο πολύ, γιατί η παρουσίαση δεν αποτελεί αντικείμενο της, διαχειρίσιμης, της ε, διατηρήσιμης διαχείρισης των δασών. Μπορεί βέβαια να ε, αναφερθούμε σε αυτά στη συζήτηση αργότερα, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να υποθεί τώρα είναι ότι στη στρατηγική 2020 τα δάση είναι ένας βασικός στόχος και για τα δάση, ο στόχος για το 2020 είναι να διασφαλίσουμε και να καταδείξουμε ότι όλα τα δάση θα τα διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη σύμφωνα με ε, ε, αρχές αηφόρου διατήρησης. Έχουμε λοιπόν την αηφόρο διαχείριση, την αποφυγή της απερίμωσης, αυτά είναι αρχές που ενισχύονται και έτσι η στρατηγική και τα δάση βέβαια καθ' αυτά, αλλά και με τη βοήθεια της στρατηγικής θα πρέπει να εξισορροπήσουν διάφορες βασικές λειτουργίες, να ανταποκριθούν στη ζήτηση και να παράσχουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων και να αποτελέσουν και βάση τη... για ανταγωνιστικότητα σε όλη την αξιακή αλυσίδα και να συμβάλλουν στις... Ε, ε, στην οικονομία βιολογικής βάσης. Στη στρατηγική έχω, ε, έχουμε αναδείξει 8 τομείς προτεραιότητας. Θα τους αναφέρω εν τάχη για να σας δώσουμε μια ιδέα για το αντικείμενό μας. Καταρχήν έχουμε το βασικό κεφάλαιο του συντονισμού και της επικοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που τονίζουμε ιδιαίτερα γιατί θεωρήσαμε ότι περισσότερη ενημέρωση και καλύτερη επικοινωνία θα βοηθούσαν πολύ το βασικό τομέα. Ένα άλλο σημαντικό είναι η συμβολή για μεγάλους κοινωνικούς στόχους. Και τι εννοώ εδώ. Πρόκειται για τα δάση ειδωμένα μέσα από μια συνολική ε, προοπτική, υποστήριξη αγροτικών κοινωνιών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της διατηρησιμότητας, προστασία δασών, ε, βελτίωση οικοσυστημικών υπηρεσιών και βελτίωση της γνωστικής βάσης. Πολύ σημαντικό και αυτό. Χρειαζόμαστε ε, καλύτερες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των δασών, όπως και περισσότερη έρευνα και καινοτομία. Σε αυτή την ανακοίνωση θα έχετε ήδη προσέξει ότι δεν υπάρχει προ... μελλοντικό πρόγραμμα δράσης για τα δάση, έτσι αποφασίστηκε, αλλά μας ενδιαφέρει να οικοδομήσουμε πάνω σε στρατηγικούς προσανατολισμούς για κάθε τομέα προτεραιότητας που παρέθεσα εντάχει πριν από λίγο, για να έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε πολύ γρήγορα το έργο μας, δηλαδή η δασική στρατηγική να αρχίσει να ε, ε, εφαρμόζεται. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να εξετάσουν τις αρχές και τους στόχους της στρατηγικής μας όταν καθορίζουν και αποφασίζουν και εφαρμόζουν τα δικά τους προγράμματα δράσης και τα εθνικά δασικά προγράμματα. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να επιτύχουμε με τη στρατηγική μας αυτή. Τώρα, τα κριτήρια για τη διατηρήσιμη διαχείριση των δασών είναι κλειδί για την επιτυχία της στρατηγικής μας. Και είναι σημαντικό, και το είπα ήδη αυτό, πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, κριτήρια αντικειμενικά και ορατά που να ε, εφαρμόζονται στην δασική βιομάζα. Χρειάζεται λοιπόν καθορισμός κριτηρίων και μετά η συζήτηση θα ε, εμβαθύνει στα κριτήρια ε, δεν θα πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά να τον εξυγχρονίσουμε. Τέλος, για τους πόρους, αυτή η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα τεκτενόμενα στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής, όπου τα δάση είναι αντικείμενα πιθανής ε, χρηματοδότησης και περιμένουμε τον κανονισμό που βελτιώθηκε για την ανάπτυξη της υπαίθρου, γιατί μας δίνει τώρα περισσότερες δυνατότητες να βοηθήσουμε τα δάση να αναπτυχθούν, όπως και οι δασικές δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν πιο εύκολα. Αυτό που δεν άλλαξε βέβαια είναι ότι αν ε, δούμε τη χρηματοδότηση στα πλαίσια της ανάπτυξης της ε, υπαίθρου θα πρέπει οι δικαιούχοι να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται τα δάση σύμφωνα με τις ε, αρχές ε, αηφόρου διαχείρισης των δασών. Υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι πόροι. Υπάρχουν, όπως σας είπα, έξι επίτροποι. Έξι επίτροποι υπέγραψαν και πρέπει να συμμετέχουν στη δασική στρατηγική. Υπάρχει το Life Συν, υπάρχει το Ταμείο Συνοχής και τα σχετικά προγράμματα, τα διαρθρωτικά ταμεία, ο Horizon 2020 με τη νέα δυνατότητα των συμπράξεων για καινοτομία στην Ευρώπη, οι πολιτικές για την ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Εδώ έχουμε και τα, το Red Plus, το FLECT Ε, ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ στα πλαίσια των συζητήσεών μας και πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις αυτές ε, βασίζονταν σε εισρωή και συνεισφορές από τα κράτη-μέλη και υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά και ε, στη συμβολή των εμπλεκομένων. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, γιατί υποστηριχθήκαμε πάρα πολύ και είχαμε και πολύ στιβαρές πρωτοβουλίες από τους εμπλεκομένους. Θα γνωρίζετε ίσως ότι έχουμε ένα μέσο διακυβέρνησης θα λέγαμε που είναι η ε, επιτροπή, ε, Δασική Επιτροπή ε, Καθοδήγησης. Η, το ανακοίνωση αναφέρει τη βελτίωση της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και να εξετάσει πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε συνοχή και συντονισμό των ε, πολιτικών που αφορούν, έχουν συνάφεια με τη δασική πολιτική. Επίσης, θέλουμε όπου χρειάζεται βελτίωση των ε, συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι θα ευγνώμων για την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων μέσα από την Επιτροπή για τα δάση με παρουσία των εμπλεκομένων που παρουσιάζουν τις απόψεις τους και έχουμε και Συμβουλευτική Επιτροπή για βιομηχανίες με βάση τα δάση. Βέβαια, δεν ξεχάσαμε κι άλλους τομείς που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον και θα έπρεπε να συζητηθούν και να καλυφθούν. Θα αναφέρω ορισμένα θέματα πρόληψη δασικών πυρκαγιών, καταπολέμηση νόσων, ζυζανίων, ε, πρόθεση ε, διατηρήσιμης ξυλίας, διαπεριφερειακή συνεργασία. Όλα αυτά είναι συνιστώσεις που θα εξεταστούν, γιατί αυτή είναι ρητή επιθυμία αρκετών κρατών μελών και έχουν καταγραφεί. Και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εμείς ήδη παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο παράλληλα με την παρουσίαση της στρατηγικής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε παράλληλη παρουσίαση και τώρα έχουμε ομάδα εργασία του Συμβουλίου για να διατυπωθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η συζήτηση έχει προχωρήσει σημαντικά. Έχουμε προχωρήσει πέρα από το 50% και είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψε με τα κράτη-μέλη. Και τώρα έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη στρατηγική μας και σε εσά ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και θα δούμε, περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα λάβετε και εσείς σχετικά με τον περαιτέρω χειρισμό της στρατηγικής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια τελευταία λέξη τώρα. Ε, έχουμε αρχίσει άμεσα το έργο της ε, υλοποίησης. Ε, υπάρχει μια πρώτη συνάντηση της ε, μόνιμης επιτροπής για τώρα το Δεκέμβρη για να δούμε πώς θα καταπιαστούμε με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν και κάναμε ανταλλαγή απόψεων ολοκληρω... και χθες μάλιστα η Κοπακοσέκα και άλλοι μας, συζήτησαν, μας κάλεσαν να συζητήσουμε με τους εμπλεκομένους ε, λεπτομερέστερα τη στρατηγική μας. Και τέλος, ευχηστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι χρειάζεται μια ε, αναθεώρηση, επανεξέταση αναθεώρηση της στρατηγικής μέχρι το 2018 για να αξιολογηθεί η ε, πρακτική εφαρμογή υλοποίηση της στρατηγικής. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Μάρκους Χόλτσερ. Η Ελίζαμπεθ Κόσιντζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μάρκους Χόλτσερ για την παρουσίαση της στρατηγικής που την περιμέναμε τόσο καιρό. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας να ε, ολοκληρώσουμε την έκθεση στα, πριν ολοκληρωθεί η θητεία του Κοινοβουλίου. Γιατί η δασική στρατηγική από το 1998 έπρεπε να τύχει επανεπεξεργασίας. Εδώ στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Γεωργίας υπάρχει μια γενική αποδοχή ότι τα δάση είναι σημαντικά για τα οικοσυστήματα και αποτελούν και πηγή ευημερίας και απασχόληση στην Ήπεθρο, αν γίνεται σωστή διαχείριση αξιοποίηση. Μια διαχείριση διατηρήσιμη είναι πολύ σημαντική και πρέπει να περιλαμβάνεται στη δασική στρατηγική ε, ως βασικό θέμα. Θα πρέπει επίσης, ε, χαιρετίζουμε την ε, ανανέωση αυτή της δασικής στρατηγικής και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Άγκρη για την ολιστική προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Η δασική στρατηγική μέχρι τώρα ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών και ε, είμαι βεβαία ότι η επικουρικότητα πρέπει να διατηρηθεί. Οι στρατηγικές λοιπόν επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ καλά και να πρέπει να υπάρχει επίσης μια, ένα όραμα για το συνολικό τομέα, μακροπρόθεσμο όραμα. Δεν πρόκειται μόνο για ευρωπαϊκή δαστική στρατηγική σημειωτέων, αλλά ξεπερνάει και τα ευρωπαϊκά σύνορα, διότι ε, το εμπόριο με δασικό υλικό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων εδώ για την Ευρώπη και μας, πρέπει να μας ενδιαφέρει να έχουμε τα κατάλληλα πρότυπα και να έχουμε και τις ε, διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή της δασικής πολιτικής. Ε, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και τους ε, ε, διατηρήσιμους πόρους. Η χρήση των δασικών πόρων πρέπει να γίνεται με τρόπο αηφόρο, διασυρίσιμο. Η πιστοποίηση της διατηρησιμότητας θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί έργο των κρατών μελών και υπάρχουν καλά κριτήρια ε, και δείκτες αηφορίας και διατηρησιμότητας. Η ανάπτυξη νέων κριτηρίων διατηρησιμότητας είναι ένα ε, κρίσιμο θέμα και στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις για τις αλλαγές χρήσης γης και δασοκομείας. Ε, δεν υπάρχει ενιαίο και όριμο σύστημα το οποίο να μπορεί να εφαρμόζεται στα 28 κράτη-μέλη μας όμως ακόμη. Τώρα, ε, δεσμευτικά προγράμματα για τη δασική διαχείριση. Εδώ υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Μια ευρωπαϊκή υποχρέωση θα ήταν άσκοπη γραφειοκρατία και θα ήταν και μέτρο δυσανάλογο. Πολλές επιχειρήσεις λόγω του γραφειοκρατικού φόρτου ε, ε, παρετούνται από τη διαχείριση κάποιων ε, δασικών περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Ε, αν χρειαστεί να παρέμβουμε στα δεδομένα των κρατών μελών, αυτό νομίζω θα ήταν υπερβολικό. Χρειάζονται ισοδύναμα προγράμματα που να μπορούν να τίθενται σε ισχύ. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό και επίμαχο θέμα ε, είναι το, η αρχή αυτή η κασκά του καταράκτη. Ε, που θα πρέπει να έχει θετικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε μεταξύ άλλων να ξεφύγουμε και από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η αρχή αυτή όμως είναι υπερβολική και ξεπερνάει και το στόχο της. Η αποτελεσματικότητα των πόρων μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς άμεση πρόσβαση στην αγορά. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε ήδη ε, είναι η μόνιμη Επιτροπή Γεωργίας, Γεωργικής Έρευνας, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ως συμβουλευτικό όργανο και είναι σημαντικό το τομέα να τον συμπεριλαμβάνουμε πάντοτε στην ε, ε, εξέταση της πολιτικής μας και όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, να παρεμβαίνουν. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα δεδομένης της ε, συνολικής προσέγγισης που θέλουμε. Ευχαριστούμε, Ελίζαμπεθ. Γιώχανσον και μετά Χόισλινγκ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση που κάνατε της νέας στρατηγικής για τα δάση. Πρέπει να σας πω πως και εγώ χαιρετίζω την προσπάθεια που γίνεται. Με βρίσκει σύμφωνο η στρατηγική και για τη δασοκομεία η περιγραφή που κάνατε πρέπει να σας πω πως είναι ένας κλάδος στον οποίο είναι πολύ δραστήρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου επηρεάζουμε ε, και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Έχει να κάνει και με τη βιομηχανική πολιτική τική και με την πολιτική έρευνα και βέβαια εν ώψη του Horizon 2020 καλό είναι να ακολουθούμε αυτή την ολιστική προσέγγιση την οποία και εσείς έχετε επιλέξει. Η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλυψε πολλά από τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα και κυρίως μας ικανοποιεί το ότι βλέπουμε μια νέα ε, στρατηγική. Έχουν συμβεί πάρα πολλά σε σχέση με την τελευταία μας ε, συνάντηση και νομίζω πως ο κλάδος της ε, δασοκομείας μπορεί να προσφέρει σε μία ανανέωση του περιβάλλοντος και να προσφέρει επίσης και στην παραγωγή ενέργειας. Η επαφή που έχω με τον κόσμο της υλοτομίας με οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το δάσος μόνο ως πρώτη ύλη, είτε για ενέργεια, είτε για ε, κατασκευές, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως έχει τη σημασία της πρώτη ύλης για πάρα πολλούς παραγωγικούς κλάδους στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται και από την υφαντουργία. Άρα λοιπόν είδαμε στο κομία και ο τρόπος που θα την χειριστούμε μπορεί να μας δώσει μια πιο βιώσιμη πρώτη ύλη για τη βιομηχανική παραγωγή ε, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο βιώσιμη η παραγωγή από το βαμβάκι, το οποίο ε, περνάει από μεγάλη χημική επεξεργασία πριν μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πολλά έχουν γίνει λοιπόν και πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα. Αν δούμε τι κάνει μια χώρα όπως η Σουηδία, στην οποία έχουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ε, περιφέρειες και αν δείτε το πώς χρησιμοποιούμε εκεί τι δασοκομεία και πόσο βιώσιμη είναι και στην κεντρική Σουηδία και στην ε, βόρεια Σουηδία, θα καταλάβετε πως πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη. Και όπως πολύ σωστά λένε οι συνάδελφοι, θα πρέπει θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό εθνικής, ευρωπαϊκής και τοπικής στρατηγικής και να δούμε ε, και πόσο θα φέρουν τμήμα της ευθύνης και οι οικονομικοί φορείς. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος καλύπτει και το κεντρικό εθνικό επίπεδο, αλλά και το περιφερειακό επίπεδο για να διαχειριστούν τέτοιου είδους ε, πόρους φυσικούς πόρους. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να προκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών στη διαδικασία χάραξης στρατηγικής για τα δάση. Μια άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει για τα υπόλοιπα τμήματα της πρότασης, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και αργότερα. Πάντως, ε, καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή, την αντιμετωπίζουμε πολύ θετικά και θα γίνουν και οι κατάλληλες συζητήσει για να χαράξουμε πλέον μια στρατηγική, μια και η δασοκομεία μας επιτρέπει να πετύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον. Άρα λοιπόν με χαρά αναμένω τις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε για τη στρατηγική για τα δάση. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Χόισλιν και μετά ο κύριο Σολενίτσα. Ευχαριστώ πολύ που συζητούμε το θέμα των δασών και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει κοινή στρατηγική και την προσαρμόζει. Για να είμαι ειλικρινής όμως δεν είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι πιστεύω γιατί τα δάση είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα πολλών δέντρων. Αν το δούμε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα δε, έχουμε ε, μεγάλη διαφορετικότητα και θα πρέπει και με διαφορετικό τρόπο να χειριστούμε τις ιδιαιτερότητες. Σε πολλές νότιες ευρωπαϊκές χώρες ε, έχουμε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών που κάθε χρόνο καταστρέφουν πολλά δάση και πρέπει να ε, φροντίσουμε για την αναγέννηση του δάσους ε, ούτως ώστε να αποκατασταθούν οι περιοχές αυτές. Κάθε χρόνο Έχουμε πυρκαγιές, αλλά μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν βλέπω. Επίσης, σε πολλές περιοχές έχουμε πρόβλημα αγωνιστικών χρήσεων. Ιδιαίτερα σε περιφέρειες αξιοποίησης υπερβολικής. Ε, εκεί ε, είμαστε υπερβολικοί. Η ξυλία είναι σημαντική, αλλά πολλές φορές φτάνουμε σε ορισμένα όρια, όπου εκεί πρέπει να πούμε ότι η σύγκρουση που υπάρχει ε, μεταξύ της ανάγκης προστασίας της φύσης και της εκμετάλλευσης πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Σε πολλές περιφέρειες έχουμε φτάσει στα όρια μας όπου μπορεί να διατρέξει κίνδυνο η διατηρησιμότητα. Στη δική μου περιοχή ε, τώρα η θέρμανση πολλών κατοικιών γίνεται με καύση ξυλίας. Ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όπως και σε άλλες περιοχές και πολύ γρήγορα φτάνουμε σε συγκρούσεις και σε ορισμένα ε, όρια σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτή και σύγκρουση με άλλους τομείς. Πρέπει να επιληθούν λοιπόν αυτές οι συγκρούσεις. Θα ήθελα τέλος να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης για διάφορα είδη δασών στην Ευρώπη και να υπάρχουν και ενιαία πρότυπα ε, με βάση τα οποία θα μπορέσουμε να ορίσουμε και να εφαρμόζουμε τα κριτήρια αηφοερίας... να αναπτύξουμε πρότυπα στην Ευρώπη ώστε από κοινού να πούμε αυτή είναι διατηρήσιμη ε, δασική ε, δασοκομεία ε, και να συμφωνήσουμε σε αυτά. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι, ακόμα και αν η δασική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ε, ορίσουμε από κοινού κριτήρια ε, βιωσιμότητας των δασών στην Ευρώπη και διατηρησιμότητάς τους. Για να ενισχύσουμε και κάποιους, κάποιους θεσμούς, θεσμικά όργανα, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο πότερος στόχος. Αν δούμε ότι τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικά, για να ενισχυθούν πρέπει να έχουν και ένα συγκεκριμένο στόχο. Ε, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε γενικές συζητήσεις χωρίς να υπάρχει αρκετή πρακτική δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρτίν, ο κύριος Ολενίτσα και μετά ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Και εγώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και αυτή την εισαγωγή στη στρατηγική για το 2020. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που γίνονται για τα δάση στα κράτη-μέλη. Δεν απαιτούμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια λύση που θα μπορέσει να, εφαρμοστεί ενιαία και ομοιογενώ σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι αδύνατο για πολλού και διάφορους λόγου. Καταρχήν δεν έχουμε κοινή πολιτική για τα δάση. Και σε χώρες μέλη με πολύ διαφορετικό τρόπο εφαρμόζεται η δασική πολιτική. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, τα δάση εμπίπτουν στην κρατική ιδιοκτησία, ενώ στη, σε πολλές ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ιδιοκτήτες των δασών μπορεί να είναι ιδιώτες ε, ή ιδρύματα ή άλλοι φορείς. Πάντως είναι σημαντικός ο συντονισμός, γιατί όταν μιλούμε για τα δάση θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η αύξηση τη δασική επιφάνεια στην Ευρώπη μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να μα αποφέρει. Καταρχήν περιορίζονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, άρα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και ένα σημαντικό άλλο πλεονέκτημα της ε, αναδάσωσης και της ε, επέκτασης των δασικών περιοχών είναι το θέμα της απασχόλησης. Πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεων εργασίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άμεση σχέση με τα δάση. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτό. Οπότε στα πλαίσια αυτά, ορίζοντας 2020, θα μπορούσε να προβλέψει και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με τη χρήση και νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε ε, στα πλαίσια των, της ε, προσπάθειας αντιμετώπισης των απειλών για τα δάση, όπως είναι οι πυρκαγιές στα δάση ή άλλων ε, τραγικών γεγονότων, καλό θα ήταν να εγκρίνουμε νέα μέτρα και να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες για να προστατεύσουμε τα δάση από τις πυρκαγιές, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό και το πρόγραμμα στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής, γιατί στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα προβλέπουμε και άμεσες ενισχύσεις για την αναδάσωση σε ιδιώτες και επίσης προβλέπουμε κάποιες δραστηριότητες για την ε, ανάπλαση και την αναδάσωση μετά από σημαντικές θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασφάλειας των δασών. Αυτό το, το έχουμε επιχειρήσει ήδη για τις ε, αρρώσιμες καλλιέργειες και για τις ε, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Έχουμε λοιπόν ε, και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες πολύ σημαντικούς, αλλά δεν έχουμε και οικονομικούς παράγοντες, γιατί τα δάση είναι πραγματικά πηγή σημαντικής πρώτης ύλης της ξυλίας, που αξιοποιείται ιδιαίτερα σε πολλούς τομείς. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι ο οικολογικός παράγοντας. Οπότε θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλες εκτάσεις που σήμερα καλλιεργούνται, είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά στο μέλλον καλό θα ήταν να είναι ε, δάση, δασικές εκτάσεις για, για οικονομικούς λόγους, για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για περιβαλλοντικούς, για οικολογικούς λόγους καλό θα ήταν ένα τμήμα των γεωργικών εκτάσεων να μετατραπούν σε δασικές. Άλλωστε, μερικές φορές έχουμε και χρησιμοποιητές ε, μεγάλες εκτάσεις, ε, είτε εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Οπότε, καλό θα ήταν ε, αυτές οι εκτάσεις εγκαταλελειμμένες να αναδασωθούν και στο μέλλον να γίνουν δάση. Γιατί σήμερα τέτοιου είδου ανεξέλεγκτε εκτάσεις έχουμε πολλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόκειται σε διάβρωση. Είναι κρίμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για βιωσιμότητα όταν μιλάμε για τα δάση. Και υπάρχει ένα δέντρο στη χώρα μου που πια δεν είναι δημόσιο. Είναι ένα είδος ιτιάς το οποίο πάσχει από μια ασθένεια που έφτασε στη χώρα μας από την Ευρώπη που θα εξαφανίσει το δέντρο αυτό από, την από, την... από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα στη δική μου εκμετάλλευση είδα τα δέντρα που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια. Βέβαια, εδώ βρίσκω πως είναι που μας προσφέρεται μια ελπίδα και ξέρω πως εάν κανείς χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει γενετικά τροποποιημένα αυτό το δέντρο μπορεί να καταλήξει σε ποικιλίε οι οποίες είναι ανθεκτικές αυτή την ασθένεια. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο με συγχωρείτε, θα μας πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω λόμπι να κάνουμε κάτι διαφορετικό ε, επειδή ε, είναι γενετικά τροποποιημένα τα δέντρα. Ähm, ναι. Καλό είναι να έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική για την ε, δασική οικονομία, τη δασοκομεία, γιατί η γεωργία και η δασοκομεία είναι σημαντική και για την οικονομία και για τη βελτίωση του κλίματος. Η δασική οικονομία και η δασοκομεία είναι πολύ σημαντική εδώ και γι' αυτό θα πρέπει να μην βλέπουμε γεωργία και δασοκομεία ανταγωνιστικά. Ο συνάδελφος Χόρσλινγκ μίλησε για την χρήση, την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση. Σε πολλές περιφέρειες, κυρίως ορεινές στην Ευρώπη, έχουμε υποεκμετάλλευση των δασών. Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Διότι η εκμετάλλευση αυτών των δασών ε, δεν αποδίδει εύκολα και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, τα δάση αυτά δεν συμβάλλουν όπως θα μπορούσαν, γιατί άμα ένα δάσος δεν ε, αξιοποιείται, ε, το ίδιο διοξίδιο του άνθρακα όπως προσλαμβάνει. Γιατί αυτό είναι μια κυκλική διαδικασία. ενώ αν χρησιμοποιηθεί ε, για υλοτόμηση και λοιπά, τότε ε, επηρεάζεται θετικά η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Ε, στη δική μου περιφέρεια, τα τελευταία 15 χρόνια, είχαμε αναπτύξει ένα καλό σύστημα για την αξιοποίηση των δασών και για την ενεργειακή κάλυψη θέρμανση κοινοτήτων και είχαμε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΚΑΠ δεύτερο πυλώνα ε, για την υλοτόμηση. Η συμβολή από το δεύτερο πυλώνα θα έπρεπε να εξυπηρετεί και όντως εξυπηρέτησε την προηγούμενη επταετία ώστε να μπορούν να, ε, οι ιδιοκτήτες των δασών να χρησιμοποιούν την ξυλία. Τα τελευταία 7 χρόνια ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε αμφισβητήσει το σύστημα αυτό όμως ε, και τώρα στην τελευταία προγραμματική περίοδο σκέπτεται να το απαλείψει. Καλό είναι όμως να υπάρξει ενημέρωση εδώ και να ξέρει η δεξιά τυπή η αριστερά. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ωραία προγράμματα και όταν πρόκειται ε, για την ε, βελτίωση της χρήσης ξυλίας σε μια δύσκολη περιοχή ε, να δημιουργούνται προσκόμματα. Ένα άλλο θέμα που ανέφερε ο συνάδελφος Χόσλινγκ αφορά την αποφυγή καταστροφής των δασών από δασικές πυρκαγιές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια ως επιτοπλίστων για την ε, αποκατάσταση των καταστροφών από πυρκαγιές. Δεν ξέρω ε, αν το έχετε σκεφτεί, γιατί έχει γραφτεί πολύ συχνά ότι οι πυρκαγιές, κυρίως στα νότιοευρωπαϊκά κράτη, είναι εμπρισμοί ε, με συγκεκριμένο σκοπό βραχυπρόθεσμη χρήση της γης. Και αυτό δεν εντάσσεται στην πολιτική προστασία των δασών. Αν υπάρχουν τέτοιες πρακτικές δεν μπορούμε να ε, παρεμβαίνουμε και να υποστηρίζουμε ακόμα περισσότερο με ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα έπρεπε η ευθύνη να αναλυφθεί από εκείνους που πρέπει ε, ε, στα κράτη-μέλη όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο των εμπρισμών. Ε, πρέπει να είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι δεν θα αποζημιώνουμε τις ε, πυρκαγιές εμπρισμούς με κοινοτικά κονδύλια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Λουίς Καπόλα Σάντος είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να χαιρετήσω την ανακοίνωσή της, αλλά θέλω να είμαι και κάπως ρεαλιστής. Το έγγραφο είναι καλό, εμπεριστατωμένο, συγκροτημένο και πιστεύω ότι θα τύχει γενικής αποδοχής. Αλλά φοβάμαι ότι δεν έχει πρακτικές ε, συνέπειες. Γιατί ως όργανο συντονισμού αυτό που προτείνεται είναι η διατήρηση της ε, μόνιμης δασικής επιτροπής και διατήρηση των ε, συμβουλευτικών επιτροπών για τα δάση, για τα ενδιατήματα και την ομάδα εργασίας για την Natura 2000. Οπότε προτείνεται η υφιστάμενη διάρθρωση συντονισμού. Σε ό,τι αφορά τα μέσα πολιτικής. Έχουμε τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα ισχύσει παρόμοιος προϋπολογισμός, αλλά είναι κυρίως ε, εκούσια μέτρα, προαιρετικά για τα κράτη-μέλη. Διαρωτώ με λοιπόν αν απλώς έχουμε εδώ μια φιλοσοφική συζήτηση, γιατί τη στιγμή που ξεκινάει η συζήτηση για μια πιθανή ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση, έχουμε ε, τα κράτη που ολοκληρώνουν τα προγράμματά τους για την αγροτική ανάπτυξη. Και θα αρχίσουν να, να αυτά τα προγράμματα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα συμπεριληφθούν ε, οι προτάσεις της ανακοίνωσης στα προγράμματα αυτά. Οπότε είναι λίγο ρεαλιστικό, να, ε, μη ρεαλιστικό να έχουμε αυτή τη συζήτηση τώρα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα έμπρακτης εφαρμογής όλων αυτών των συστάσεων. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση και να δούμε πώς ε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει υπόψη την ε, έγκριση των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που αυτόν τον καιρό συζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας ε, για την συμμετοχή στη συζήτηση και να σας υπενθυμίσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων Ομάδων δεν έχει δώσει ακόμη την έγκρισή της ε, για την ε, σύνταξη τρεχούσης κοινοβουλευτικής θητείας μιας έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για την ε, νέα δασική πολιτική ή στρατηγική. Οπότε χωρίς τέτοια έγκριση δεν προλάβουμε εμείς στην κοινοβουλευτική αυτή θητεία μας να συντάξουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Πάντως ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξαναδώσω το λόγο στον Διευθυντή Μάρκους Χόλτσερ για τα συμπεράσματα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος και μάλλον θα επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, το θέμα των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ακολουθεί από τότε που άρχισε η συζήτηση. Όντως είναι περίπλοκο το θέμα, πολύ. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ειδικά στο πρόγραμμα ανάπτυξης υπαίθρου υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αλλά και προγράμματα αποκατάστασης. Δεν σημαίνει αυτό ότι δίνουμε τα χρήματα χωρίς να εξασφαλίζουμε αξία για τους Ευρωπαίους. Ε, δρούμε προληπτικά θα έλεγα για διάφορους λόγους. Όχι μόνο προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές αλλά προλαμβάνουμε και καταστάσεις μετά την πυρκαγιά, ε, μια κατάσταση καταστροφική για την βιοπικιλότητα και αποτρέπουμε και πολλές αρνητικές επιπτώσεις έτσι. Αυτό το μονοπάτι το ακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό και αποδείχθηκε με όλους βέβαια τους περιορισμούς που υπάρχουν ε, από τα κράτη-μέλη, για τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες της Κομισιόν αποδείχθηκε ότι βρήκαμε έναν τρόπο αντιμετώπισης. Και είπα και προηγουμένως κατά την παρουσίαση ότι ε, αυτό το έχουμε αναδείξει σημαντικό θέμα της στρατηγικής μας. Τώρα για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις νόσους, γιατί ετέθη ένα ερώτημα εδώ. Βεβαίως γνωρίζουμε το πρόβλημα με το συγκεκριμένο δέντρο και μας απασχολεί η ανάπτυξη. Μπορεί όμως να υπάρχουν δυνατότητες να καταπολεμήσουμε τις νόσους ε, για αυτό το δέντρο, το φράξο. Είναι σημαντικό για μας και το έχουμε εντοπίσει όχι μόνο το πρόβλημα του δέντρου φράξεως αλλά τους επιβλαβείς, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις νόσους γενικότερα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τη στρατηγική μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας βέβαια. Τώρα, για τη φιλοσοφική συζήτηση, εντόπισα μια αναφορά που έγινε. Δεν είναι η δασική στρατηγική, δεν είναι φιλοσοφικό ζήτημα. Μπορεί να μην είναι για τον Α ή τον Β αρκετά συγκεκριμένη και λεπτομερής, αλλά με τα κράτη-μέλη, με τους εμπλεκομένους, καταλήξαμε κάπου. Και ε, ε, εδώ παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Εδώ και δύο χρόνια συνεχίζεται η συζήτηση αυτή. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, η στρατηγική να ε, είναι υπερβολικά καθυστερημένη γιατί στην προπαρασκευαστική φάση όπου τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες ε, γνώριζαν τα πορίσματα των συζητήσεων και μπορούσαν να ε, λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά όταν εκπονούν τα προγράμματά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε τη στρατηγική μας Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο κατάφερε να ε, εντάξει αυτό το θέμα ε, στις εργασίες του για φέτος. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας μας διάταξης για να προλάβουμε να ανταλλάξουμε και τις χριστουγεννιάτικες ευχές. Σημείο 8 λοιπόν, παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κοινοτικού Γραφείου για τις φοιτικές ποικιλίε. Θα μας κάνει την παρουσίαση ο κύριος Μάρτιν Έκβατ, που είναι ο πρόεδρος αυτού του Κοινοτικού Γραφείου για τις φοιτικές ποικιλίε. Θα γίνει λοιπόν η παρουσίαση των δραστηριοτήτων αυτών, γιατί στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά δικαιώματα για τις φοιτικές ποικιλίε. η κατάσταση πια έχει αλλάξει όπως γνωρίζετε και ιδιαίτερα ο κανονισμός που προτείνεται για το αναπαραγωγικό φυτικό υλικό περιλαμβάνει νέες αρμοδιότητες για το κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών. Ενώ ο κανονισμός για τα για, τις, για το σύστημα δικαιωμάτων για τις φυτικές ποικιλίε θα υποστεί αναθεώρηση στο έγκυς μέλλον. Ε, φαίνεται ότι λίγοι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν τις ε, δραστηριότητες ε, του σημαντικού αυτού γραφείου. Στο παρελθόν είχαμε και ελάχιστη επικοινωνία με το γραφείο αυτό. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την εκπόνηση μελέτης για τις δημοσιονομικές πτυχές της λειτουργίας των αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν να δώσω το λόγο στον Διευθυντή, στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Γραφείου για τις Φυτικές Ποικιλίες, τον κύριο Έκβατ. Σας ακούμε κύριε Έκβατ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρων για την πρόσκληση να κάνω την παρουσίαση αυτή. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, κατά το παρελθόν δεν υπήρχαν πολλές επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που έρχομαι να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώτη φορά το γραφείο παρουσιάζει τις δραστηριότητες του στην Επιτροπή αυτή από ότου άρχισε το 1995. Ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε πιο στενά. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπήρχαν ε, τυπικά θέματα που έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη για την ομοθεσία δηλαδή. Τώρα έχουμε τον κανονισμό PRM, όπου όπως είπε και ο πρόεδρος ε, προβλέπονται περισσότερα καθήκοντα για το Κοινοτικό Γραφείο Φοιτικών Ποικιλιών και το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί επί της νομοθετικής πρότασης. Έχουμε και τον ιδρυτικό μας κανονισμό που ε, αξιολογήθηκε πριν από ε, λίγα χρόνια και επίσης θα αναθεωρηθεί νομικά. Και εσείς θα συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, είμαι βέβαιος. Υποθέτω μάλλον. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, έγινε μία μελέτη για τους αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς. Ένα είναι το γραφείο, είναι καλή μελέτη και παρουσιάζει τα επίμαχα θέματα είναι ενδιαφέρον και καλό ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τα οικονομικά μας. Είναι όμως και καλή ευκαιρία για μένα σήμερα να παρουσιάσω ορισμένες από τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες. Γενικά η καινοτομία είναι θέμα κλειδί για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε ένα οικονομικό κλίμα που είναι όλο και πιο περιπλοκό. Πιο συγκεκριμένα η καινοτομία στα φυτά είναι σημαντική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που πρέπει να ε, έχουν τρόφιμα και, λιγότερο, περιορισμένο αριθμό εκτάσεων ή περιοριζόμενων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ποιότητα για τους καταναλωτές, να καταπολεμήσουμε επιβλαβείς οργανισμούς νόσους και υπάρχουν και πολλές προκλήσεις σχετικά με τις ποικιλίε που θα πρέπει να είναι ε, αηφόροι και βιώσιμες στο περιβάλλον. Ε, υπάρχει καινοτομία ε, σε σχέση με τα βάση που ήταν το προηγούμενο θέμα που παρακολούθησα στη συζήτησή σας ε, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να γίνουν νέες ποικιλίε δασικές που θα ανθίστανται σε πυρκαγιές κλπ. Η προστασία λοιπόν, η φυτοπροστασία είναι πολύ σημαντική και ένας οργανισμός αποτελεσματικός από το χρηματοδοτούμενο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Ε, εμάς ε, τα οικονομικά μας είναι διαφανή, ελέγχονται παρκώς και είναι λογικό το κοινοτικό γραφείο να αναλάβει νέα καθήκοντα στον τομέα των φυτικών ποικιλιών. Ε, με ενημέρωσαν ότι έχω δεκάλεπτο για την παρουσίαση. Μπορεί να λίγο παραπάνω για να κάνω μια παρουσίαση του οργανισμού, να δώσω στατιστικά συνεχεία, να μιλήσω για τα οικονομικά μας, τα νέα καθήκοντα μετά το σχέδιο κανονισμού για το αναπαραγωγικό φυτικό υλικό, αξιολόγηση του συστήματος και κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Καταρχήν το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε με βάση κανονισμού του Συμβουλίου χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου το 1994 και τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ε, χορηγήθηκαν στα πλαίσια αυτού του συστήματος και ισχύουν στο έδαφος των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, υπάρχει με τα εθνικά συστήματα των 24 κρατών μελών της Ένωσης που έχουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας για τις φοιτικές ποικιλίε και θα επιλέξει ο ετών αν θέλει να τύχει εθνικής προστασίας ή ενωσιακής προστασίας, όλη την επικράτεια της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα ευθυγραμμίζεται με την Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φοιητικών Ποικιλιών, την UPOV, είναι σύμβαση του 1991 και είναι υπόδειγμα για το ενωσιακό σύστημα. 24 από τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης είναι μέλη της ε, σύμβασης UPOV η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως μέλος της UPOV ως ε, διακυβερνητικού οργανισμού. Ε, λειτουργεί ως οργανισμός ομπρέλα σε όλο τον κόσμο. Το ενωσιακό σύστημα για την ε, προστασία των φυτικών πηγικυλιών είναι ένα σύστημα ιδιαίτερο ε, ε, οι δημιουργοί της ποικιλία εξαιρούνται, όλες οι ποικιλίε, ε, προστατευόμενες ή όχι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή για περαιτέρω έρευνα από τους δημιουργούς των νέων ποικιλιών, χωρίς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την αμοιβή τους ή λόγω νομικών θεμάτων. Υπάρχουν και γεωργικές εξαιρέσεις, δηλαδή οι γεωργοί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιούν στις εκμεταλλεύσεις τους προστατευόμενες ποικιλίε. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούν να προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνία ή φοιτικέ ποικιλίε με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ευρεσιτεχνιών και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τι Ευρεσιτεχνίε και τα διπλώματα που χορηγούνται σε βιοτεχνολογικέ εφευρέσει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιε γκρίζε ζώνε και στι ευρεσιτεχνίε μια συζήτηση που συνεχίζεται και θα τη γνωρίζετε. Τώρα, για το κοινοτικό γραφείο. Καταρχήν ο οργανισμός έχει μια δήλωση αποστολής που δηλώνει ότι θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία στις φυτικές ποικιλίε με υψηλή ποιότητα σε επεξεργασία των αιτήσεων ε, για δικαιώματα ε, στις φυτικές ε, με λογικό κόστος ενώ ε, δίνουμε κατευθυντήριες ε, πολιτικές γραμμές και υποστήριξη στην άσκηση των δικαιωμάτων για τους εμπλεκομένους. Υπάρχει το γραφείο από το 1995 με έδρα στην Ανζέ στη Γαλλία. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του γραφείου ορίζονται από, διορίζονται από το Συμβούλιο και έχουμε 45 μέλη προσωπικό από 12 εθνικότητες. Είμαστε από τους μικρότερους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινοτικό γραφείο ε, διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει μια επιτροπή προσφυγών, όπου μπορούν να προσφεύγουν οι πελάτες αν δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις που λαμβάνομαι. Και αν συμβαίνει αυτό, και αν δεν, ε, ε, αν δεν καλυφθούν από την Επιτροπή Προσφυγών μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Ε, συνεργαζόμεθα στενά με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιορισμένη μόνο ήταν η συνεργασία όπως σας είπα. Πολύ σημαντικό είναι ότι συνεργαζόμεθα στενά με γραφεία ε, που κάνουν τεχνικές εξετάσεις τις οποίες εμείς χρειαζόμαστε πριν λάβουμε απόφαση σχετικά με χορήγηση ή μη χορήγηση κάποιου δικαιώματος για φυτική ποικιλία. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί το κοινοτικό γραφείο και αποτελείται από εκπροσώπους των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανισμούς παρατηρητές. Είναι η μη χορηγηση καποιου δικαιωματος για φοιτικη ποικιλια το διοικητικο συμβουλιο παρακολουθει το κοινοτικο γραφειο και αποτελειται αρχή του γραφείου και όπως είδατε στη μελέτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό του Κοινοτικού Γραφείου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με ποια γραφεία θα συνεργαστούμε ε, στα κράτη-μέλη, ποια γραφεία μπορούν να αναλάβουν την διεξαγωγή τεχνικών εξετάσεων γιατί πρέπει να πληρούν ποιοτικά κριτήρια και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν πληρούν τα γραφεία τα κριτήρια αυτά. Επίσης, ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο τα τεχνικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για να κρίνουμε αν είναι σταθερή, διακριτή ε, η ποικιλία και ε, αυτά τα πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται και στη γεωργία και στον φυτικό τομέα όταν γίνεται αίτηση για ε, έγκριση στην αγορά. Είμαστε 45 στο γραφείο όπως σας είπα, δεν έχουμε δημιουργήσει δική μας τεχνική υποδομή, χρησιμοποιούμε τα γραφεία των κρατών μελών και ε, αυτά ε, λειτουργούν ε, παντού για να φροντίσουμε ότι όλες οι περιβαλλοντικές συνθήκες λαμβάνονται υπόψη όταν γίνονται κάποιες, ε, κάποια τεστ, κάποιες δοκιμές. Από την αρχή της ίδρυσής μας ε, λάβαμε περίπου 48.000 αιτήσει και το 2010 αρχίσαμε σύστημα αιτήσεων online. Τρία χρόνια αργότερα τώρα έχουμε το 65% των αιτήσεων με το σύστημα online. Ε, χορηγήσαμε περισσότερους από 36.000 τίτλους, πάνω από 21.500 είναι ενισχύ και έχουμε 1.800 διαφορετικά είδη. Έχουμε πολύ τεχνογνωσία, ε, ανάγκη ε, και τη βρίσκουμε στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν είναι μικρά τα γράμματα και εδώ χωρίζομαι τις αιτήσει τομέα καλλιέργειας και βλέπετε ότι οπότε τότε που άρχισε να λειτουργεί το γραφείο ο τομέας των καλοπιστικών είναι ο μεγαλύτερος. Από εκεί έρχονται οι περισσότερες αιτήσει. Περίπου το 60% των αιτήσεων έρχονται από το τομέα των καλοπιστικών. Έχουμε και τα γεωργικά είδη που είναι περίπου 23-24%, μετά έχουμε τα κυπευτικά 12% και φρούτα 6% των αιτήσεων. Και είδαμε σχεδόν σταθερή τάση αύξησης αριθμητικά των αιτήσεων κατέτος θέτος Έχουμε ήδη σπάσει το ρεκόρ, δεν φαίνεται στη διαφάνεια περάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Δηλαδή έχουμε περίπου 3.200 αιτήσει για νέε ποικιλίε από ευρωπαϊκές και άλλες εταιρείες πέρσι. Εδώ βλέπετε μία κατανομή των αιτήσεων αναχώρα, από ποιες χώρες ελάβαμε πέρυσι και βλέπετε ότι η Ολλανδία είναι κατά πολύ η πρώτη χώρα στην υποβολή αιτήσεων. Μετά έχουμε τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία. Φαίνονται στη διαφάνεια οι χώρες από τις οποίες ε, λάβαμε αιτήσει. Επίσης ε, παίρνουμε και από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρώτη είναι, πρώτος είναι η Ευρωπαϊκή οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ολλανδία, Ιαπωνία, το 20% των ε, τήσεων προέρχονται από μη, χώρες ε, μη κράτη-μέλη και το 80% από τα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ ότι παίρνουμε ε, τήσεις από όλο τον κόσμο. Αυτά πολύ σύντομα ε, οι δραστηριότητες του γραφείου. Τώρα, για τα οικονομικά μας ορισμένα πράγματα λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε. Ανέλησε λοιπόν η μελέτη τον καθορισμό των τελών, την αντιμετώπιση δημοσιονομικών πλεονασμάτων και τη διαδικασία απαλλαγής. Καταρχήν, στο σύστημά μας η Κομισιόν αποφασίζει για το επίπεδο των τελών που θα καταβάλουν οι ετούντες όταν υποβάλουν την αίτησή τους. Ε, βασίζεται η απόφαση σε πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου. Εκεί στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εμείς είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός, όπως σας είπα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο αφενός, από την άλλη θα πρέπει να εξισορροπούμε δύο αντιρροπούμενους στόχους. Ο πρώτος είναι να διασφαλίσουμε την συνέχεια των ε, λειτουργιών μας, Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετά οικονομικά μέσα για να διεξάγουμε τι δραστηριότητέ μα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη χρήματα, αν μα τελειώσουν. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πάντοτε θα έχουμε επαρκή κονδύλια για τι δραστηριότητέ μα. Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα χρημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρούμε το απόθεμά μα σε ένα λογικό επίπεδο. Και αυτό καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο, ένας λόγος, ένας λόγος που είναι δύσκολο αυτό είναι ότι ο οργανισμός μας διέπεται από τη ζήτηση, δηλαδή στην αρχή του χρόνου δεν ξέρουμε πόσες ζητήσεις θα παραλάβουμε, πόσους, πόσοι τίτλοι θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχύοι και γι' αυτό δεν είναι τόσο προφανές Ε, και τόσο εύκολο να έχουμε έναν ισορροπημένο ισολογισμό από χρόνο σε χρόνο, θα πρέπει να δούμε μια περίοδο που θα καλύπτει 2 με 5 χρόνια για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ισορροπημένο ε, προϋπολογισμό. Ε, εδώ μία ένδειξη για τα τέλη που εισπράττουμε, ένα τέλος ε, αίτησης που θα καταβληθεί από τον ετούντα πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε τον φακελό του. Υπάρχει το τέλος της εξέτασης ανάλογα με την καλλιέργεια, το είδος. Υπάρχει ένα διοικητικό τέλος σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη έκθεση σε ένα κράτος μέλος και μπορεί να την αναλάβουμε αυτή, να την πάρουμε εμείς. Αυτό στοιχίζει 250 και μετά έχουμε ένα ετήσιο τέλος το οποίο τώρα ανέρχεται σε 300 ευρώ. Πρέπει κανείς να τα καταβάλει αυτά τα χρήματα ε, για να είναι ενισχύει ο τίτλος. Από 1η Ιανουαρίου φέτος μειώθηκε από 900 σε 650 το τέλος ε, αίτησης και από το 2014 το ετήσιο τέλος θα μειωθεί και αυτό. Και γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί αυξάνεται το απόθεμά μας και πρέπει να το ξανακατεβάσουμε στα επίπεδα που πρέπει. Τα τελευταία χρόνια, με βάση τους λογαριασμούς μας, βλέπουμε πλεόνασμα και το 11 και το 12. Ήταν ο προϋπολογισμός περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ και η αύξηση, τα κέρδη, για να το πω έτσι, τα καθαρά ήταν 1,5 εκατομμύριο. Από τότε που μειώσαμε, από την 1η Ιανουαρίου φέτος, τρέχοντος έτους δηλαδή το τέλος ε, για την αίτηση, τώρα θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα 0,5 μισό εκατομμύριο, 500.000 και του χρόνου, όταν το ετήσιο τέλος θα μειωθεί, θα έχουμε έλλειμμα στον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να ε, πάμε το απόθεμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί στο απόθεμα ήταν πολλά τα χρήματα για τα τέλη και το 2011 αποφασίσαμε να περάσουμε αυτό το μέτρο για να έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα μέχρι το 2014. Βλέπετε ότι το 2013 θα είμαστε περίπου στις 500.000 και λίγο παραπάνω και αυτό θα αντιστραφεί και θα μας δώσει αρνητικό αποτέλεσμα ε, της τάξης του 1 εκατομμυρίου το χρόνο για να κατέβει το απόθεμα στα σωστά επίπεδα, εκεί που πρέπει. Τώρα, τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Είπα ότι μειώσαμε τα τέλη Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι υπέρ αυτής της ιδέας της μείωσης των τελών. Στηρίζουν τις προσπάθειές μας να μειώσουμε τα τέλη, αν και οι αιτήσει ε, στα κράτη-μέλη μπορούν να χάσουν λίγο από εκεί, γιατί θα είναι λιγότερο δαπανηρό να ζητήσει κανείς προστασία ε, σε νοσιακό επίπεδο από το να κάνει πολλές αιτήσει σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης. Εμείς επενδύουμε το πλεόνασμα με βάση μια πολιτική επενδύσεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ε, εξετάζεται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ε, αυτό ήταν ένα... Η απαλλαγή είναι ένα θέμα που εξετάστηκε από τη μελέτη επίσης. Πρέπει να πω ότι για τη διαδικασία της απαλλαγής ε, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι ανεξάρτητος φορέας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται βέβαια από τα κράτη-μέλη και κατανοούν πολύ καλά τα συστήματα και ξέρουν τα μέσα και τα έξω του οργανισμού. Βασίζεται η απαλλαγή σε μια γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και έχουμε και εσωτερικούς ελέγχους θεσμοθετημένους Λαμβανομένων όλων τούτων υπόψη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το κοινοτικό γραφείο ελέγχεται, αξιολογείται και εξετάζεται περισσότερο από τους περισσότερους ε, οργανισμούς σε ό,τι αφορά τη δαπάνη κάθε ευρώ. Τώρα, για τον ε, κανονισμό ε, PRM για το πολλαπλασιαστικό υλικό, το φυτικό υλικό. Εδώ τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι ικανοποιημένα που έχει αναλάβει το ρόλο ε, το γραφείο. Ε, θα έχουμε δηλαδή εμείς το Μητρό των Ποικιλιών σε, Ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χειριζόμεθα τις αιτήσει ε, για κάποια είδη ε, χρειάζεται εξουσιοδότηση από τα κράτη-μέλη σε, κάποια, σε κάποιες ποικιλίε. χρειάζεται εξουσιοδότηση από τα κράτη-μέλη ε, προς το κοινοτικό γραφείο και εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις μέχρι να συμφωνήσουν σε όλο αυτό τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Εμείς ε, παρέχουμε συμβουλές στα κράτη-μέλη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς των ποικιλιών και έχουμε και έλεγχο σε μεγάλο βαθμό των γραφείων εξέτασης. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει η τροπολογία του ιδρυτικού κανονισμού. Υπήρξε μια αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε το 2011 από μια εταιρεία που ανέλαβε εξουσιοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέληξε ότι το σύστημα λειτουργεί καλά συνολικά και οι εμπλεκόμενοι είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα και θέλουν να το διατηρήσουν με την τρέχουσα μορφή του αν και θα χρειαστούν κάποιες προσαρμογές προσεκτικής στόχευσης. Δεν περιμένουμε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν αναλάβει το ε, ρόλο της η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το Κοινοτικό Γραφείο Φοιτικών Ποικιλιών ε, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ε, τη υποβολή των αιτήσεων μπορούν να πάνε σε ένα γραφείο για να υποβάλουν την αίτηση αντί να πηγαίνουν στη χώρα του. Είναι λιγότερο ο διοικητικό φόρτο για τι εθνικέ αρχέ, εμεί αναλαμβάνουμε διοικητικά, όχι τεχνικά καθήκοντα. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοτικού Γραφείου και τα κράτη-μέλη σε τεχνικό επίπεδο και η προστασία παρέχεται συνολικά σε λογικές τιμές. Επίσης, η δημοσιονομική διαχείριση, το είπα ήδη, είναι υγιής και ε, η λογική είναι νέα καθήκοντα να, ε, να τίθεται σε ένα ενωσιακό οργανισμό. Έχουμε τώρα πάνω από 12 χρόνια εμπειρία ε, και ο κανονισμός για το πολλαπλασιαστικό υλικό ε, τώρα θα εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη αλλά ε, ε, ε, παρακολουθείται από το κοινοτικό γραφείο. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσω. Λαμπρά, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε του Κοινοτικού Γραφείου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση που έγινε από το γραφείο σας, από τον και κύριο Έκβατ ε, για τις δραστηριότητε αυτού του πολύ σημαντικού κοινοτικού γραφείου. Κανένας όμως συνάδελφος δεν ζήτησε το λόγο, δεν ξέρω. Θέλει κανείς το λόγο? Ο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Έχω κρατήσει σημειώσεις για τον οργανισμό που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Καλή ιδέα. Μακάρι να ίσχυε και για άλλους, γιατί έχουμε πολλούς. Καλό θα ήταν το επιχειρηματικό μοντέλο να το παρουσιάσουμε και σε άλλους ε, στο γεωργικό τομέα. Στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου θα γίνει η αξιολόγηση και θα συζητηθεί πάλι ο βασικός κανονισμός. Ε, σε αυτό το τομέα γνωρίζετε και εσείς ότι ε, υπάρχουν προβλήματα, ε, προστασία του εδάφους Χρειαζόμαστε εδώ να λύσουμε θέματα όπως το, δημιουργία... Έχουμε το πρόβλημα ε, στην κτηνοτροφία. Ε, υπάρχουν όμως ε, πολλές προσπάθειες να παρακαμφθούν τα συστήματα ε, μια τεχνική διαδικασία μπορεί να αποκτήσει ε, δίπλωμα έβρεση τεχνίας και μετά να περάσουν και σε ποικιλίε. Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια νομικά τρίκ που πρέπει να τα αποφύγουμε. Δεν θέλουμε δημιουργία μονοπωλίων, πρέπει να υπάρχει ελευθερία για τους γεωργούς. Τέλος, να προσέξουμε στον ε, οργανισμό σας, όλα να γίνονται νομότυπα και κάποιες πολιτικές αρχές που έχουμε και που ε, είναι αποδεκτές από όλους, αυτές οι αρχές λοιπόν να συνεχίσουν να υλοποιούνται. Ε, εδώ πάντα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ πολιτικών και πρακτικών εφαρμογών. Καλό είναι λοιπόν να συνεχίσουμε την επαφή και τις συζητήσεις μεταξύ μας, γιατί ο ρόλος σας είναι σημαντικός ως γραφείο και, στην, ε, και είναι σημαντικός και για τη γεωργία, αλλά και για τα συμφέροντα των ε, γεωργών. Ευχαριστώ, Πέτερο. Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου για την παρουσίαση αυτή που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και νομίζω πως μας ε, παρουσιάσατε πολλά στοιχεία τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε. Αυτό το οποίο με εντυπωσίωσε ήταν ε, κάτι που είπατε, ότι υπάρχει λιγότερη υγεία η οποία πρέπει να παράγει περισσότερα τρόφιμα για περισσότερους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση για την ΚΑΠ. δεν είναι μόνο τα ε, φυσικά στοιχεία όπως ο καιρός, οι εποχές που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Είχαμε τη μεγάλη ξηρασία πέρυσι στη ΣΥΠΑ που εκτείναξε τις τιμές και βλέπουμε διαφορετικές τελείως οδείες φέτος. Άρα λοιπόν δύο χρονιές ποτέ δεν μοιάζουν. Ίσως αυτό είναι και το πλεονέκτημα το ότι δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε το τι καιρό θα κάνει, γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε πώς να συμφωνήσουν όλοι για το τι καιρό πρέπει να κάνει. Καλό είναι λοιπόν που δεν έχουμε εμείς και αυτή την ευθύνη. Τώρα, εσείς είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι ιδρυθήκατε την ε, δεκαετία του 90 και είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας να κάνετε μία παρουσίαση. Υπάρχει κάτι λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα γιατί όταν δημιουργείτε νέες ποικιλίε ή καταγράφετε νέες ποικιλίε που είναι πιο ανθεκτικές ε, στις ασθένειες για παράδειγμα Τι σημαίνει για σας ε, το γενετικά τροποποιημένο. Προηγουμένως ο κύριος Άγνιου μίλησε για το πρόβλημα της μελιάς στην παρουσίαση που έκανε. Ε, εσείς κάνετε κάτι γιατί μπορεί βέβαια να διαφωνούμε και στην ίδια την Επιτροπή για το θέμα αυτό και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, στην Ευρώπη δεν ε, έχουμε καταλήξει μια κοινή πορεία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα εξαφανιστεί στο μέλλον. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει παραμένοντας η μοναδική Ήπειρος η οποία δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Jim. E Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Καπούλας και μετά θα ακούσουμε την απάντηση του Πρόεδρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Γραφείου για την ενημέρωση που μας έκανε. Τη βρήκα πολύ χρήσιμη. Γιατί έτσι εξοικειωθήκαμε με ένα σημαντικό τμήμα του έργου του Κοινοτικού Γραφείου που πραγματικά δεν γνωρίζαμε. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτού του Κοινοτικού Γραφείου μόνο το γεγονό ότι μία απόφαση που λαμβάνεται εκεί εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη δημιουργεί μια τεράστια πλούστευση για του ε, οικονομικού τελεστέ. Θα ήθελα εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα λοιπόν να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση που μα κάνατε. Ευχαριστώ και θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο του Κοινοτικού Γραφείου για τι φοιτικές ποικιλίε, τον κύριο Άρκο, για την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση για το γενετικός τροποποιημένο υλικό. Θα έλεγα ότι ευτυχώς μάλλον εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Για να αποφευστεί κατά πόσο ένα γενετικός τροποποιημένος οργανισμός μπορεί να καλλιεργηθεί και να τεθεί σε εμπορία, αποφασίζουν ε, οι Εθνικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι το δικό μας γραφείο. Αν μια ποικιλία είναι γενετικώς τροποποιημένη ή όχι, δεν είναι θέμα που μας απασχολεί. Εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη νέα ποικιλία, εμείς μπορούμε να δώσουμε τίτλο. Και το αν ε, μπορεί να πολιθεί, όχι να τεθεί σε πώληση, θα αποφασίσουν άλλες αρχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, θα ήθελα να πω ότι λίγες ποικιλίε γενετικώς τροποποιημένες κυκλοφορούν σε εμάς σε σχέση με, με άλλες χώρες. Εμείς ξεκινήσαμε το σύστημα με λιγότερο από 100 αιτήσει για γενετικώς τροποποιημένες ουσίες και μόνο ούτε καν 10 δεν έχουν πάρει τον τίτλο την άδεια κυρίως γιατί δεν μπορούν να τεθούν σε ε, εμπορία αυτές ε, οι ποικιλίε ως γενετικώς τροποποιημένες, παρόλο που τη χάνουν προστασίας. Εμένα η κατάσταση με ικανοποιεί πλήρως. Και στο μέλλον φυσικά το γραφείο θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Τώρα με ρωτήσατε και για τη συνεργασία του γραφείου μας με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Είπα στην παρουσίασή μου ότι έχουμε τακτική, πολύ τακτική και στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, που είναι η αρμόδια διεύθυνση της, Γενικής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε στενή συνεργασία για τα θέματα αυτά με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε στο μέλλον να εντείνουμε αυτή τη συνεργασία θα πρέπει μη τι άλλο να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ ευχαρίστω θα, θα έλθουμε να σα κάνουμε παρουσιάσει για πολλέ πτυχέ του έργου και των δραστηριοτήτων μα. Γιατί στο μέλλον η ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε νομοθετικό επίπεδο για τα θέματα αυτά θα είναι πολύ πιο σημαντική. Είναι ευπρόσδεκτες αυτές οι εξελίξεις και εμείς ε, προσβλέπουμε σε εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με το Κοινοβούλιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους ε, στη δεξίωση που έχουμε ετοιμάσει εκτός της αίθουσας, μπροστά στην αίθουσα. Όλοι είστε προσκεκλημένοι, ευρωβουλευτές, βοηθοί, υπάλληλοι για να ανταλλάξουμε χριστουγεννιάτικες ευχές και να κάνουμε και μια πρόποση για τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ θερμά και ραντεβού στην επόμενη συνεδρία στον Ιανουάριο.